Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ακρόαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μας είναι καθοδόν. Αποφασίσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ακρόαση παρόλα αυτά. Να πω λίγα λόγια εν είδη εισαγωγής και έπειτα ως εισηγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα κάνω και κάποια προκαταρκτικά σχόλια για την ακρόαση. Ο τίτλος είναι «Ο χάρτης ως το σημείο αναφοράς για τη μελλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή της». Συγγνώμη, ο αντίκτυπο του χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης». Όπως θα γνωρίζετε, η Υποτροπή ΛΥΜΠΕ αυτής εξ αρχής θεωρεί το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το θεμέλιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και των σχετικών πολιτικών. Υπό αυτήν την προοπτική, από το 2000, ο χάρτης ήταν σημείο αναφοράς και για το Ευρωκοινοβούλιο και για τις εκθέσεις μας για την διάδοση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Το 2005 και το 2007 αντιστοίχω, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ οργάνωσε δύο ακροασει συναντώντα τι ύψιτε αρχέ τη Ευρώπη ε, που είναι υπεύθυνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, καθώ και εκπροσώπου από τα εθνικά συνταγματικά τμήματα, δικαστήρια και του ενδιαφερομένου από την κοινωνία των πολιτών μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και της ίδιας της ε, χάρτας, η οποία έγινε υποχρεωτική σημασία, καταλαβαίνουμε τώρα τον πραγματικό αντίκτυπο αυτού του κειμένου. Στο πόσο επηρεάζει δηλαδή την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την υλοποίησή της στα κράτη-μέλη. Ο στόχος αυτής της τρίτης ακρόασής μας, κατά σειρά, είναι να λάβουμε κάποια καθοδήγηση για τις προοπτικές που ανοίγονται με το νέο νομικό πλαίσιο, να δούμε πώς διαμορφώνεται η μελλοντική νομοθεσία και να αποτιμήσουμε ξανά το κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με τα θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Η ακρόασή μας θα, θα συναποτελείται από τρία μέρη. Σήμερα θα έχουμε το πρώτο μέρος και θα επικεντρωθούμε στο θέμα του χάρτη ω σημείο αναφορά για τη μελλοντική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εφαρμογή τη σε εθνικό επίπεδο. Το δεύτερο τμήμα τη ακρόαση θα αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπω θεσπίστηκε από τα ανώτατα δικαστήρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αύριο το πρωί θα έχουμε ένα τρίτο μέρο όπου θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη και το χώρο τους, τη στατηγική της Επιτροπής και την άποψη του ακαδημαϊκού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών και των Εθνικών Ινστιτούτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κάθε τμήμα της ακρόασης θα περιλαμβάνει και ένα μέρος συζήτησης ερωταπαντήσεων, πράγμα που θα γίνει και σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί δηλαδή. Η συμμετέχοντες μπορούν να ζητούν το λόγο βεβαίως για την συζήτηση και παρακαλούνται να ενημερώνουν το Προεδρείο επισημένοντας το όνομά τους και τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν στο φυλάδιο το οποίο θα μοιραστεί στην αίθουσα. Οι διάφοροι προσκεκλημένοι μας, οι οποίοι θα παρέμβουν στη συζήτηση, θα πρέπει να μιλήσουν 8 με 10 λεπτά, ώστε να παραμείνουμε εντό χρονοδιαγράμματος. Και ήθελα να παρακαλέσω όσους θα ζητήσουν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, να παραμείνουν σε ένα σύντομο πλαίσιο δύο λεπτών, ώστε να σεβαστούμε το πρόγραμμα που προβλέπετε για την απογευματινή μας ακρόαση και την αυριανή. Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και ως εισηγήτρια για την έκθεση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνω τώρα το ρόλο και το καθήκον να σας παρουσιάσω κάποιες εναρκτήριες παρατηρήσεις, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε και αργότερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα νέο ρυθμό, ένα νέο δρόμο που ανοίγεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για έναν δρόμο που ανοίγεται μετά την Λισαβόνα, μετά το Δεκέμβριο του 2009 δηλαδή. Έχουμε πλέον το δεσμευτικό χάρτη και έχουμε υποχρέωση να τηρούμε τα, τις υποχρεώσεις της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα νέο όργανο που ασχολείται με το θέμα αυτό, έναν νέο θεσμικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίτροπο επεφορτισμένο με τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, η οποία θέλει να παρακολουθεί συστηματικά και να επιβάλλει και τις απαιτήσει των Ευρωπαίων πολιτών σε όλη αυτή την προσπάθεια και έχουμε και τον οργανισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να παρακολουθεί και να υποβάλει εκθέσεις για τα θέματα της υλοποίησης της, του χάρτη. Αυτά είναι τα κοινοτικά όργανα. Επίσης υπάρχουν τα δικαστήρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Αυτό που βλέπουμε εδώ να διαμορφώνεται είναι ένας κατάλογος με θεσμικά όργανα νομικώς δεσμευτικά εργαλεία και αφού θεσπίστηκαν ε, οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορούμε να έχουμε εδώ, το θέμα είναι πώς θα τις αξιοποιήσουμε, τι χρήση θα έχουν, πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα εργαλεία, οι μηχανισμοί και τα θεσμικά όργανα που έχουν ε, θεσπιστεί. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να γίνει το σύστημα αυτό να λειτουργεί ομαλά, να αρχίσει να λειτουργεί ομαλά και να βεβαιωθούμε ότι τα θεσμικά όργανα θα εφαρμόζουν τις νομικές υποχρεώσεις που έχουν προκύψει. Επίσης, θεωρούμε ότι θα είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την τήρηση των υποχρεώσεων του χάρτη από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την χρήση του κοινοτικού δικαίου και τον χάρτη. Και όταν αυτό βεβαίως είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε την υλοποίηση του χάρτη όποτε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνουν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να τηρούν και τις υποχρεώσεις του χάρτη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία παραμένει συνεπής με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να το κάνουν ε, σε συνεργασία και με τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Η υλοποίηση και σε επίπεδο κοινοτικό και σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει, όπως προείπα, να εξασφαλίζει τη συμβατότητα με το χάρτη. Ξεκινώντας από την κοινοτική νομοθεσία και καταλήγοντας στην εθνική νομοθεσία θα μεταφέρει κοινοτικέ πράξεις. Αυτές είναι οι απαιτήσει που προκύπτουν από το χάρτη, από την ύπαρξη του χάρτη. Τώρα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τους καλύτερους τρόπους και μέσα που διαθέτουμε από αυτή τη σκοπιά, όποτε στο μέλλον διαδούμε να απαιτείται κάτι σε σχέση με την υλοποίηση του χάρτη. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο όπου η Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, με μένα την ίδια υπεύθυνο εισηγήτρια ετοιμάζει μία έκθεση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν ως εισηγήτρια πιστεύω ότι τώρα είναι ευθύνη μας να δούμε τα υπάρχοντα θεσμικά μέσα και να δούμε ποιος κάνει τι στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και επίσης τι ρόλο πρέπει να διδραματίσει κάθε θεσμικό όργανο και πώς όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε. Να συνεργαστούμε και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο επίπεδο των κρατών μελών. Να δούμε δηλαδή πώς τα δικαστήρια μπορούν μεταξύ τους να συνεργαστούν και τι μπορούν να κάνουν από κοινού για να αποφευχθούν διπλές προσπάθειες, περιττές προσπάθειες. Να δούμε δηλαδή πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τους διεθνείς οργανισμούς, στα θέματα που επηρεάζονται από την εφαρμογή του χάρτη. Όπως τα διαφορετικά σώματα του ΟΗΕ, ή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχει η πληθώρα ευρωπης υπαρχει εδώ, τα οποία πρέπει να γύρουμε και να συζητήσουμε. Νομίζω στην έκθεση αυτή που ετοιμάζουμε τώρα στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να καλύψουμε τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε εδώ σήμερα για να μας βοηθήσετε να δούμε τι κάνει το κάθε θεσμικό όργανο, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός και πώς θα μπορούσε εδώ να δράσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω ότι αν όλα τα θεσμικά όργανα του Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένου διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο σε αυτό το νέο αρχιτεκτόνημα, με αυτό το πολύ σύγχρονο χάρτη, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτές οι προσδοκίες είναι πολύ ψηλέ αφού δημιουργήσαμε και θεσπίσαμε την ίδρυση τόσων θεσμικών μηχανισμών. Συνάδελφοι, φίλε και φίλοι, αυτές ήταν οι ιδέες που ήθελα να σας υποβάλω προκειμένου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Επιτρέψτε μου τώρα να ζητήσω από τον κύριο Πίτερ Χάστινγκς, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, να πάρει το λόγο για να μας παρουσιάσει όσα έχει να μας πει. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι ίσως σύμπτωση που προγραμματίστηκε ομιλία για τον Ευρωπαίο Επόπτη της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Στην ακρόαση αυτή, όπου θα ακούσουμε διάφορες παρεμβάσεις από εκπροσώπους διαφόρων οργάνων, από την Ισπανική Προεδρία, από όλα τα όργανα που ασχολούνται με την προστασία των δικαιωμάτων της Χάρτας των Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για την επιρροή που θα έχει η Χάρτα στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Γι' αυτό και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δραστηριοποιείται όλος ιδιαιτέρως ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σας ευχαριστώ. Αυτό συνδέεται και με το πρόγραμμα της Στοχόλμης που εγκρίθηκε στα τέλη του περασμένου έτους. Εκεί προεξάρχοντα ρόλο έχει η συλλογή, η ανταλλαγή και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητα εργαλεία για την εκπόνηση κοινοτική πολιτική στον τομέα του ασύλου, της ε, αστυνομική συνεργασία, της μετανάστευση και της εσωτερικής ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο τονίζεται η ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείριση των πληροφοριών. Τα καλά νέα είναι ότι πέρα από την ε, ανταλλαγή πληροφοριών, ως αντιστάθμισμα αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και άρα καλωσορίζω τη βαρύτητα που αποδίδουμε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διαχείριση των Προσωπικών Πληροφοριών. Και φυσικά καλωσορίζω το ρόλο που έχει η προστασία των δεδομένων γενικότερα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Η σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων πλέον είναι δεσμευτική μέσα από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και επαναλαμβάνεται αυτή η σημασία ε, σε διάφορα σημεία της συνθήκης. Υπάρχει μια διάταξη στην οποία θα επανέλθω, άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από το άρθρο 8, ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δίπλα στο άρθρο 7 σχετικά με την ιδιωτικότητα των πληροφοριών. Μέσα στο άρθρο 8 επιβεβαιώνεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρεται και στο άρθρο 16. Έτσι, οι πολίτες αντικειμενικός πώς έχουν ένα δικαίωμα το οποίο μπορούν να επικαλεστούν και ενώπιον των δικαστηρίων. Βέβαια, υπολείπεται να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των δικαστηρίων, εάν γίνει κάποια σχετική προσφυγή και επιπροσθέτω υπάρχει και το άρθρο 6.2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει σαφής ερήτρη για την πρόσβαση, για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προσχώρηση που πλέον είναι υποχρεωτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε τη βαρύτητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τώρα στο άρθρο 16 της συνθήκης αναφέρεται ότι η θεμελιώδης αξία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων επιβεβαιώνεται και τονίζεται. Αναλύοντας αυτή τη διάταξη, διακρίνουμε σαφώς πως τα βασικά στοιχεία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ε, είναι, ας το πούμε, θέσφατα πλέον, διότι αναγνωρίζονται στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο. Υπάρχει αντικειμενικό δικαίωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι σαφής η διατύπωση στο άρθρο 16 και υπάρχει πλέον νομική βάση. Δηλαδή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων οπωσδήποτε πρέπει να έχει ένα νομικό έρισμα, μια νομική βάση. Αναγνωρίζεται επίσης η αρχή του περιορισμού λόγω σκοπού της χρήσης των πληροφοριών, το δικαίωμα πρόσβασης ε, στα δεδομένα κάποιου. Το η αρχή επίσης της εποπτείας από μια μερόληπτη αρχή. Όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία αναγνωρίζονται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χώρος της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ως εκ τούτου δεν μπορεί να οικοδομηθεί εάν ε, δεν υπάρχει πλήρης σεβασμό του δικαιώματος προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 8 και κατόπιν στο δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο. Γι' αυτό όταν ε, υπάρχουν ε, σχέδια νομοθετημάτων και κατόπιν εγκρίνονται, σας παραπέμπω στον κατάλογο των σημείων δράση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι εντυπωσιακό. Έχει γίνει μια απογραφή και υπάρχει ε, και στην ιστοσελίδα μας. Ε, δηλαδή ό,τι σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών ε, δεδομένων. Ποιοι θα εμπλέκονται για την εξακρίβωση του σεβασμού όλων αυτών των επιμέρου στοιχείων κατοχυρώντα έτσι την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην ιστοσελίδα μου ανεβάζαμε αυτό το κατάλογο στις αρχές του τρέχοντος μήνα αλλά και σε εθνικό επίπεδο θα είναι εφαρμοστές αυτές οι διατάξεις όταν εφαρμόζεται η νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο και στο άρθρο 51 της χάρτας ε, σαφώς προσδιορίζεται ότι οι εθνικές ε, αρχές οφείλουν να τηρούν αυτή τη διάταξη επιπλέον θα πρέπει να ερμηνεύεται η χάρτα σε πλήρη συμμόρφωση με την νομολογία του δικαστηρίου ε, και στο Στρασβούργο και στο Λουξεμβούργο όλη η νομοθεσία στον χώρο της ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης, άρα και για την ανταλλαγή πληροφοριών, καλύπτονται από αυτές τις ρήτρε. Και ε, βλέπουμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτός ο νέος ρόλος των, ε, της προστασίας των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έρχονται εδώ και διάφορες ενδιαφέρουσες αποφάσεις ε, του ε, Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Η υπόθεση Χούμπερ, παραδείγματος χάρη, όπου ε, η μη διακριτική μεταχείριση λόγω εθνικότητας και εθνοτικής προέλευσης ήταν το διακύβευμα ως προς τα δημοτολόγια. Ε, ή ως προς τους ε, ε, καταλόγους για τους μετανάστες. Υπάρχει νομολογία στο Στρασβούργο σχετικά με τις βάσεις δεδομένων για τα για τους επιβάτες, η υπόθεση Μάρμπερ, μία σειρά υποθέσεων που διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο για την προετοιμασία και την εκπόνεση νομοθεσία στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το θέμα της μη διακριτικής μεταχείρισης ε, και το ε, ε, για κάποια άτομα, παραδείγματο χάρη, που υπάρχει το όνομά του σε καταλόγους για τον έλεγχο των συνόρων, πλέον δεν είναι κάτι αφηρημένο και το θεωρητικό. Σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τώρα την αναθεώρηση της ε, υφιστά, του υφιστάμενου δευτερογενούς νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών ε, δεδομένων. Είναι ένα από τα σημεία δράσης του προγράμματος της Στοκχόλμης και αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει η προστασία των δεδομένων. Από 1η Πρώτου του 2009 εξάλλου η προστασία των δεδομένων και η τήρηση των επιμένων στοιχείων κατοχυρώνται σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν μπορεί να υπάρξουν νομικά κενά. Όμως, προς το παρόν υπάρχουν για τον πρώην τρίτο πυλώνα, παραδείγματο χάρη, το ισχύον πλαίσιο δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να ισχύει βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Η απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων έχει περιορισμένο εύρο και δεν καλύπτει τι εγχώριε υποθέσει, όπω τις ονομάζουμε. Δηλαδή, όχι όταν συλλέγονται τα δεδομένα μόνο σε εθνικό επίπεδο και μετά διαβιβάζονται, αλλά σχετίζονται και με υπηκόους άλλων χωρών και άρα στη συνέχεια μπορεί στη συνέχεια να ανταλλαχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις ε, αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. Αυτή είναι μια ε, πραγματικότητα στην οποία, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και άρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό ε, το νομικό πλαίσιο. Εν κατακλείδη. Γίνεται δεσμευτική πλέον η χάρτα και προβλέπονται σημεία αναφορά για το νέο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση για την ένωμη προστασία. Αυτό προετοιμάζει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πλέον απαράδεκτο να υπάρχουν νομικά κενά και γι' αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα οριζόντιο πλήρε αποτελεσματικό πλαίσιο και Οφείλουμε επίσης να λάβουμε υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για οποιαδήποτε νέα νομοθετήματα, δυνάμει και το άρθρο 52 της ε, συνθήκης, προβλέπονται εξαιρέσεις, πλην όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και η πιθανή εξαίρεση και η ε, ακριβής εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητα είναι θέματα που σίγουρα θα απασχολήσουν μελλοντικά το Κοινοβούλιο ε, ε και θα έχουν και μάλιστα προεξάρχοντα ρόλο. Οι εξαιρέσει ε, μπορούν να ισχύσουν μόνο όταν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και είναι πλήρως αιτιολογημένες. Αυτή ήταν η καταληκτική μου παρατήρηση. Ευχαριστούμε κύριε Χάστινγκς. Τώρα θα ε, περάσουμε στην πρώτη συζήτηση. Έχουμε δύο βουλευτές που θα ήθελαν ε, το λόγο και κατόπιν ε, μπορείτε όλοι οι υπόλοιποι να ζητήσετε το λόγο αν το επιθυμείτε. Σηκώστε απλώς το χέρι σας και οι συνάδελφοι θα σας φέρουν τον κατάλογο για να εγγραφείτε. Ο κύριος Κοέλιο θα πάρει πρώτος τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια θερμά για αυτή την πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια στον Πίτερ Χάστινγκς για την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση που έκανε. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι η προστασία των δεδομένων είναι ένα σαφές παράδειγμα για το πώς η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει μεγάλη σπουδαιότητα, ιδιαίτερη σημασία στον χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ως φιλευρωπαϊστές που είμαστε, η Χάρτα σήμαινε ένα βήμα προς τα εμπρός δεν είμαστε στην Ευρώπη απλά μόνο των, της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Είμαστε στην Ευρώπη των πολιτών, όπου οι κοινέ μας αξίες βρίσκονται στο επίπεδο των συνθήκων και εκεί θεμελιώνονται. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα του χώρου της ελευθερίας, ελευθερίας δικαιοσύνης, και ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των απαντήσεων που θα δίνουμε στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας που πρέπει να διαφοροποιούνται από τις αρχές αυτές που είναι κοινέ σε όλους μας και έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα όταν εμπλέκεται σε διεθνείς δράσεις η Ευρώπη με διαφόρους εταίρους όχι μόνο με τις ΕΥΠΑ, ΕΕ, ώστε αυτές ε, οι ε, εταιρικές ας το πω έτσι δραστηριότητες θα πρέπει να βρίσκονται στα όρια και στα πλαίσια που καθορίζεται από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Χάρτα λοιπόν έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τον χώρο αυτό της δικαιοσύνης και ελευθερίας και όπως ανέφερε ο κύριος Πίτερ Χέστινγκς, στην ανάπτυξη όλων των κοινοτικών δράσεων πρέπει να λαμβάνετε αυτό υπόψη. Αυτή τη στιγμή άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να σεβόμαστε σε όλες τις παραμέτρους αυτή τη χάρτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Κυρία Τσίπερ, σας ευχαριστώ πρόεδρε εγώ νομίζω ότι σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση που διεξάγουμε. Λυπούμε για το ότι πολλοί συνάδελφοι δεν είναι σήμερα παρόντες, δεν μπορούν να παραστούν. Διότι πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα μας συναδέψει επί μεγάλο χρονικό διάστημα και οι συνάδελφοι με κάποιους άλλους τρόπους θα πρέπει να δώσουν συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση. Όταν κάνουμε λόγο για τη σημασία της προστασίας των δεδομένων και τη συνεργασία θεσμικών οργάνων, <clears throat> πολλές αποφάσεις δεν είναι μόνο τυπικά νομικές αλλά πρόκειται για μια πολιτική αξιολόγηση και πολιτική συζήτηση οι θεμελιώδεις αυτές αρχές δεν είναι καινούριε, αλλά έχουμε μια καινούρια στάθμιση με την ε, έγκριση και έναρξη σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Και από τις πρώτες συζητήσεις στην Ευρωβουλή καταδεικνύεται πόσες μεγάλες προσπάθειες δίνουμε για να υπάρξει η σωστή ε, θέση των κέντρων βάρους. Και επειδή εδώ πέρα από το πρόγραμμα της Στοχόλμης και πέρα από το θέμα του κατά πόσον τα δικαιώματα αυτά και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά και την την αστυνομία, διοκτικές δράσεις, αλλά και πολλούς καθημερινούς τομείς. Σε πολλούς τομείς έχουμε συζήτηση κατά πόσον οι προσωπικές μου ας το πω έτσι παράμετροι για την υγεία μου για παράδειγμα με την εισαγωγή και θέσπιση μιας κάρτας υγείας κατά πόσον αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέροντα για κάποιους που δεν θα έπρεπε κανονικά να ενδιαφέρονται για αυτά. Και υπάρχει συζήτηση για παράδειγμα ότι οι εργοδότες ενδιαφέρονται για τέτοια στοιχεία για να αξιολογούν κατά πόσον ένας μελλοντικό εργαζόμενος που θα απασχολούσαν εκείνοι θα αντιμετώπιζε κινδύνους από πλευράς υγείας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ανάλογα τα θέματα των ε, πολιτικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των πολιτών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν πρέπει αποκλειστικά να σταθμίζονται εναντί άλλων ε, τομέων. Η συζήτηση όμως έχει μια πολύ σαφή πολιτική πρόσθετη αξία. Με τη συζήτηση για τη σημασία των δεδομένων αυτών και των αρχών αυτών, μετά από μεγάλες συζητήσεις για την ενιαία εσωτερική αγορά και πολλές άλλες συζητήσεις, θέτουμε τον πολίτη ως άτομο στο επίκεντρο των προβληματισμών μας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτή τη συζήτηση, τις συζητήσεις για τις ε, επόμενες εβδομάδες. Και με ενδιαφέρει για το πώς εμείς αυτή τη διαχείριση δεδομένων, αλλά και και την ασφάλεια δεδομένων στη συζήτηση μπορούμε να οδηγηθούμε σε αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο το θέμα ποιος θα έχει πρόσβαση σε τράπεζες δεδομένων τέτοιων στοιχείων αλλά και πόσο επίκαιρα, επικαιροποιημένα θα είναι τέτοια στοιχεία. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαγράφονται θα διαγράφονται πραγματικά και δεν θα διατηρούνται. Και αυτό είναι θέμα το οποίο ανήκει στη συζήτηση και θα μας απασχολήσει κατά πόσο αυτά τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να επιληθούν και κατά πόσον από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ζητηθεί να υπάρξει αντίστοιχη δράση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Χάστινγκς να τονίσω αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Κοέλιου. Είναι πολύ σημαντικό ο ρυθμός που ήδη διαθέτουμε να διατηρηθεί. Η Επίτροπος Ρέντινγκ μας είπε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επιδίωξη της ενίας αγοράς. Και όπως είπα και εγώ στις αναρκτήριες παρατηρήσεις μου, έχουμε πλέον έναν ευρωπαϊκό χάρτη. Την πλέον σύγχρονη κωδικοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων παγκοσμίω. Είναι λοιπόν ένα άριστο θεμέλιο για να ξεκινήσουμε και να χτίσουμε κάτι προς όφελος των πολιτών. Κύριε Χάστινγκς. Έχετε το λόγο παρακαλώ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, νομίζω ότι η ιδέα των διοργανωτών ήταν να δείξουν ότι η προστασία των δεδομένων είναι ένα ιδιαίτερα εύστοχο παράδειγμα των επιπτώσεων της εφαρμογής του χάρτη στον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας Συμφωνώ απολύτως. Όμως, η σχέση είναι αμφίδρομη. Όπως έχει υπογραμμιστεί. Ο χάρτης καλύπτει περισσότερα από ό,τι απλή προστασία δεδομένων και όλα αυτά τα δικαιώματα, η μη διακριτική μεταχείριση, η ανθρωπίνη αξιοπρέπεια, η επεξεργασία των δεδομένων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης και την προετοιμασία της καινούργιας νομοθεσίας. Η άλλη προοπτική και αυτή ισχύει ότι δηλαδή η προστασία των δεδομένων δεν είναι εύστοχη μόνο, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το χώρο δικαιοσύνη, ασφάλεια και ελευθερία. Το... Ο στόχο τη Επιτροπή να υποβάλει προτάσει ω το τέλο τη φετινή χρονιά για την αναθεώρηση του υπάρχοντο νομικού πλαισίου εκφράστηκε στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος της Στοκχόλμης. Πρώτο μέρος του εγχειρήματο αυτού, θα το ξανατονίσω, είναι να καλυφθούν όλοι οι χώροι των ευρωπαϊκών πολιτικών. Από την εργασία, την υγεία, ως τις μεταφορές, την κοινωνική ασφάλεια και ούτω καθεξής. Μιλάμε εδώ για ένα εγχείρημα λοιπόν Πολύ σημαντικό. Επίση, τι προκλήσει των νέων τεχνολογιών, τη παγκοσμιοποίηση, πρέπει και αυτέ να τι αντιμετωπίσουμε. Επίση, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη οι επιπτώσει τη υλοποίηση του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η ενημερωτική στρατηγική μα και η επικοινωνιακή μα στρατηγική, έτσι όπω εξελίσσεται, θα μας προσδώσει μια μεθοδολογία ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα, τα λάθη που έχουν συμβεί τα τελευταία 5 με 10 χρόνια δεν θα επαναληφθούν. Δεν θέλουμε να βιαστούμε ούτε να κάνουμε μια σειρά από ενέργειες που μετά να αποτιμήσουμε, αλλά να προχωρούμε βήμα το βήμα. Και με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ευθύς εξ αρχής. Έτσι λοιπόν θα συμφωνούμε με κάθε τέτοια κίνηση εφόσον ακολουθείται αυτή η βασική προσέγγιση. Τώρα, μιλώντα γενικώ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, να μην ξεχνούμε ότι ο υποφορτισμένο με αυτό το θέμα επίτροπο, μάλλον επιφορτισμένο με αυτό το θέμα επίτροπο, ο επίτροπο Ρέντινγκ, έχει εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσουμε μια ε, πολιτική μηδενική ανοχή. Νομίζω ότι ίσω είναι κάπω υπερβολική αυτή η διατύπωση έτσι κι αλλιώς υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του χάρτη και της συνθήκης. Και υπάρχει μια ιδιαίτερη σημασία εδώ και για την προστασία των δεδομένων, αλλά και γενικότερα. Έτσι λοιπόν κάθε τέτοια πρωτοβουλία θα την υποστηρίξουμε. Και παρακολουθούμε πιστά την νομοθεσία κατά την εφαρμογή της. Θα είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί και προσεκτικοί, να είστε βέβαιοι. Ευχαριστούμε κύριε Χάστινγκς. Εφόσον άλλοι συνάδελφοι ή προσκεκλημένοι δεν ζήτησαν το λόγο, περνούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας ακρόασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρώπινη εξωπρέπεια και τη ανθρώπινη μάλλον εξωπρέπειες όπω θεσπίστηκε από τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τρεις ομιλίες εδώ. Και μετά από, την... από τις παρεμβάσεις αυτές θα κάνουμε την επόμενη συζήτηση. Να θυμίσω σε όσους θέλουν να πάρουν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης να συμπληρώσουν τα στοιχεία του στο φυλάδιο που θα κυκλοφορήσει. Ώστε να εγγραφούν. Ο δεύτερος ομιλητής μας Μάλλον πρώτο μα ομιλητή στο δεύτερο μέρο τη ακροασία είναι ο Ζαν-Κλοντ Μπονισό, πρόεδρο του τέταρτου τμήματο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε. Thank you, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω στα γαλλικά, αν δεν σας πειράζει, γιατί είναι πολύ ευκολότερο για μένα. παρότι ο τίτλος αυτής της συνόδου σχετίζεται με τον τρόπο που τα νότερα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατοχυρώνουν το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτρέψτε μου να μην ε, περιγράψω διεξοδικά ε, τον τρόπο με τον οποίο κατοχυρώνεται αυτή η προστασία από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό το θέμα και μου φαίνεται ότι θα παρουσίαζε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς, δεδομένου του αντικειμένου της ακροασής σας, να ε, εξετάσω ε, εξελικτικά το ζήτημα και να αναρωτηθώ ποιος είναι ο πιθανός αντίκτυπος της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εξάλλου αυτός είναι ο βασικός τίτλος της ε, σημερινής και αυριανής ακρόασης. Θα πω κάποια λόγια μόνο για το θέμα της προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το θέμα αυτό προφανώς συνδέεται με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ένα δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα θεσμικό όργανο ε, διοικητικού και συνταγματικού χαρακτήρα που εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποστολή της είναι να ελέγχει την νομιμότητα των ε, πράξεων και νομοθετημάτων των οργάνων της Ένωσης. Στα πλαίσια δε αυτού του ελέγχου καλείται προφανώς, όπως θα έκανε οποιοδήποτε εθνικό δικαιοδοτικό όργανο, καλείται λοιπόν να αποφανθεί για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα από τις δράσεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το δικαστήριο έχει επίσης ως πρωταρχική αποστολή να κατοχυρώσει την ομοιομορφία κατά την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου και κατά την εφαρμογή του δικαίου αυτή η ομοιομορφία είναι μια προϋπόθεση εκ των όνου κάνευ για την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο που οι συνθήκες δεν συμπεριλάμβαναν ένα κατάλογο δικαιωμάτων, μια απογραφή δικαιωμάτων, το δικαστήριο προσπάθησε να καλύψει αυτό το κενό μέσα από την ομολογία του. Είναι πλούσια η νομολογία αυτή και εμπνέει η εμπιστοσύνη. Για να εκπονήσει την ομολογία της στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το Δικαστήριο της Ένωσης προσέφυγε στις Γενικές Αρχές Δικαίου. Προφανώς εμπνεύστηκε από τις συνταγματικές παραδόσεις, κοινέ συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών της Ένωσης και από τις συνθήκες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες είχαν προσκορήσει τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο και βάσει ενός γνωστού τύπου απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ιδιαίτερη βαρύτητα λέω στην Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακολουθεί και εφαρμόζει την ομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου και επικαλείται όλο ένα και συχνότερα την ομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου στις αποφάσεις του. Ε, προστατεύει η νομολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. Είναι βέβαια πολύ άριθμα τα παραδείγματα. Η απόφαση Καντή, πολύ γνωστή από την 3η Σεπτεμβρίου 2008, όπου χάρη στην απόφαση του το δικαστήριο υπερασπίστηκε τα άτομα ή τις ε, ε, νομικές οντότητες που ε, καταγράφονται σε καταλόγους ε, τρομοκρατικών οργανώσεων. Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου ε, παρέπεμψε αυτό το θέμα στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου κατά την εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση του, της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων από εγκληματικές πράξεις ούτως ώστε να ε, θεσπιστούν ε, οι κανόνε καταγγελία ε, των δράσεων ξεπλήματος βρώμικου χρήματο. Στη συνέχεια το Συμβούλιο τη Επικρατεία της Γαλλία ανέπεμψε το θέμα στο δικαστηρίο για την εγκυρότητα και την νόμιμότητα της οδηγία σχετικά με τι ποσοστώσει για τα αέρια του θερμοκηπίου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα, οι ανώτατες δικαιοδοτικές αρχές ε, των κρατών μελών ε, θεώρησαν ότι κατοχυρώθηκε ε, η προστασία των δικαιωμάτων μέσω της δράσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέται κανείς λοιπόν γιατί χρειάζεται η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι αδιαμφισβήτητα χρειάζεται. Ε, στο στάδιο εξέλιξης που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στο βαθμό που έχει ευρύτατες πλέον αρμοδιότητες δεν είναι φυσιολογικό να μην υπάρχει κάπου μια δήλωση, ένας κατάλογος των δικαιωμάτων κατόπιν. Είναι οι τομείς όπου μπορεί να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στι αστικέ και ποινικέ υποθέσει και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Αυτοί οι νέοι τομεί όπου μπορεί να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσουν απαραίτητη την ύπαρξη ε, μια χάρτα ε, δικαιωμάτων. Τέλος, ε, και νομίζω στο σώμα που βρισκόμαστε οφείλουμε να το αναφέρουμε, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας γενικότερος προβληματισμός που θα καταλήξει σε μία ρητή επιβεβαίωση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, τώρα που υπάρχει η χάρτα των δικαιωμάτων πρέπει να αναρωτηθούμε ποια θέση έχει μέσα στην ένωμη τάξη της Ένωσης. Έτσι αναρωτιόμαστε ποια είναι η αξία της χάρτας, το περιεχόμενό της και ε, η όρη ερμηνείας της χάρτας αυτής. Ε, Ω προς την νομική αξία της ε, χάρτας σημειώστε παρακαλώ τρία σημεία. Πρώτον, η χάρτα έχει την αξία του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωση ε, αναγνωρίζει την ίδια νομική αξία για τη χάρτα όπως αυτή που έχουν οι ίδιες οι συνθήκες. Δεύτερον, το πεδίο εφαρμογής προσδιορίζεται πλέον. Η χάρτα είναι εφαρμοστέα σε όλες τις δημόσιες αρχές ε, ε, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα κράτη-μέλη φυσικά εφαρμόζεται όταν ε, υλοποιείται το ενωσιακό δίκαιο σε εθνικό επίπεδο και τονίζεται αποκλειστικά και μόνο όταν εφαρμόζουν τα ενωσιακά νομοθετήματα τα κράτη-μέλη. τρίτων η τάξη ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τροποποιείται με τη χάρτα, άρα και αυτό έχει θεμελιώδη σημασία, δεν μπορεί να αποτελέσει νέα νομική βάση αυτή η χάρτα. Ως προς το περιεχόμενο θα υπάρχουν τρία σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η χάρτα συμπεριλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σχεδόν που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα διάφορα πρωτόκολλα της σύμβασης αυτής που δεν πρέπει να ξεχνούμε. Έτσι, Εάν κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση, διαπιστώνουμε ότι 19 ελευθερίες και δικαιώματα ε, ε, είναι κοινά για την Χάρτα και για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Πέντε μόνο υπάρχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά όχι στη Χάρτα. Και ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε πως η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, αποδίδει συνταγματική αξία στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια της ένομης τάξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά η χάρτα υπερβαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση γιατί κατοχυρώνει και άλλα δικαιώματα που δεν προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. 31 δικαιώματα, 12 που σχετίζονται με την αλληλεγγύη και είναι στον τίτλο, στο αντίστοιχο κεφάλαιο που, για την αλληλεγγύη. 8 σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και 11 σχετίζονται με άλλα ζητήματα. Α ε, εξετάσουμε σφαιρικά το ζήτημα. Ένα μεγάλο τμήμα των κατοχυρωμένων πλέον δικαιωμάτων σχετίζονται όντω με την κατηγορία αυτή, δηλαδή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα, δεν ισχύει μάλλον αυτόματα για ολόκληρη τη χάρτα. Κάποια δικαιώματα, όπως αυτά που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, ε, έχουν ε, ε, κέρια σημασία για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ίσως όχι γενικότερα. Παραδείγματο χάρη το δικαίωμα καλή διακυβέρνηση. Είναι ε, ε, προτιμότερο να έχουμε μια εύρυθμα λειτουργούσα διοίκηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα όπως η ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα στο να ζει κάποιο σε ασφάλεια και ούτω καθεξής. Τώρα θα ήθελα να επιμείνω τονίζοντα το θέμα τη ερμηνεία τη συνθήκη. Περνώ στο τρίτο σημείο τη παρέμβασή μου. Και στο προήμιο και στο άρθρο 52 η χάρτα προβλέπει του κανόνε ε, δυνάμει των οποίων πρέπει να ερμηνεύεται. Η ίδια η χάρτα δηλαδή προσδιορίζει του κανόνε τη ερμηνεία τη. Τέσσερα σημεία θα ήθελα να παρατηρήσουμε σε αυτό το τομέα. Πρώτον, η έννοια και το πεδίο των δικαιωμάτων που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Χάρτα πρέπει να είναι πάνω μοιότυπα. Δεύτερον, ε, οι διευκρινήσεις οι επεξηγήσεις υπό την αιγίδα του Προεδρείου της Σύμβασης ε, ε, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Αυτό το λέει η χάρτα σαφώς και στο πρέμιο και στο άρθρο 52. Τρίτο στοιχείο, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ε, κοινή σταγματική παράδοση των κρατών μελών πρέπει να ερμηνεύονται και παραθέτω ε, σε αρμονικό τρόπο με τη χάρτα. Τέλος παράθεση, τέταρτο στοιχείο, ο περιορισμός των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται μέσα στη χάρτα θα πρέπει να αιτιολογείται. Είτε επειδή υπάρχει ανάγκη προστασίας ε, των ε, ελευθεριών ε, του, ή του δημοσίου συμφέροντος, είτε για λόγους καλής εύρυνης λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθημερινή βάση ή για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις κατευθυντήριες ερμηνευτικές γραμμές που είναι και κάπως αντιφατικές ομολογουμένως και προσθέσουμε και αυτή την σκοτεινή πρόταση του 6.3 ε, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που λέει ότι Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον πρόεδρο Μπαταντέρε ε, πρώην πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γαλλίας, που είχε πει και παραθέτω δεν μπορούμε παρά να δείξουμε σκεπτικισμό σε σχέση με ε, προληπτικά μέτρα που νομικώς πώς δεν έχουν κανένα νόημα. Ε, δηλαδή σε τελευταίο βαθμό τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ερμηνεύσουν αυτά που σας είπα ότι πρέπει η χάρτα να ερμηνεύεται σε αρμονία με το περιεχόμενό της. Ε, διότι αυτή η προληπτική ε, προσέγγιση είναι αντιστρόφω ανάλογη προ το νομικό περιεχόμενο και την νομική αξία τη συνθήκη. Θα ήθελα να προσθέσω τώρα ότι οι διευκρινήσει του Προεδριού είναι και αυτέ αντιφατικέ. Πρόεδρε, θα κλείσω σε δύο λεπτά ε, μιλώντα για την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπεται η προσχώρηση στο άρθρο 6 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπό τους όρους που προσδιορίζονται σαφώς από το πρωτόκολλο υπαριθμών 8 που έχει ισότιμη ε, νομική αξία όπως και η Συνθήκη. Γνωρίζετε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν τακτικές θυματικές και αγαστές σχέσεις και παρακολουθούν εκ του συνεγγύης ε, η νομολογία ε, το ένα του άλλου. Η προσχώρηση λοιπόν θέτει διάφορα ζητήματα ε, πολιτικού και τεχνικού χαρακτήρα εφόσον φυλάμε για αφηρημένε έννοιε. Ε, πρέπει όμω να μεριμνήσουμε τόσο ώστε μελλοντικά να λειτουργήσει εύρυθμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ε, διευθετήσουμε αυτά τα νομικά ζητήματα. Πρώτον, ποιο είναι το καθεστώ του πρωτογενού δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κυρίως ε, μιλώντας για τους όρους ερμηνείας του και για το ε, κομμάτι των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηθελημένα ε, δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου από τους δικαστές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, το ίδιο ισχύει για τους ε, όρους που θα κατοχυρώσουν την αρχή της επικουρικότητας και μην ξεχνάτε ότι ο έλεγχος γίνεται από το δικαστήριο ως προς την αρχή της αναλογικότητας. Είναι απαραίτητη η αρχή της αναλογικότητας και χαρακτηρίζει τις σχέσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά χρειάζεται ούτω ώστε δύο δικαστέ να μην επιλαμβάνονται μια υπόθεση ταυτόχρονα και επίση για να μπορεί το δικαστήριο πλήρω να ασκήσει την αρμοδιότητα που του αποδίδει η συνθήκη ε, κυρίως ε, να μεριμνήσει και να ε, ερμηνεύεται ομοιόμορφα το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα που θα χρειαστούμε, ούτω ώστε να επιλύσουμε αυτήν την μόνιμη ανταπάρε... στην επίλυση αντιδικιών ανάμεσα στα δύο δικαστήρια, αν ανακύψουν, που δεν έχει συμβεί, αλλά δεν είναι και απίθανο. Αυτά τα ε, στοιχεία νομίζω πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, ούτω ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα να έχουν τη θέση που τους πρέπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τη σήμερα ημέρα το 2010. Um, Σας ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Μελκιόρ, πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Βελγίου, πρόεδρος του 12ου Συνεδρίου της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Δικαστηρίων. Κύριε Μελχιόρ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο τίτλος Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Βελγίου ίσως κάποιος να τους εκπλήσει. Γιατί υπάρχουν δύο πρόεδροι για το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου, καθότε βρισκόμαστε σε μια ομοσπονδή χώρα. Στο Βέλγιο, με σύνταγμα ομοσπονδή χώρα. Τώρα, για το δεύτερο τίτλο που αφορά τον πρόεδρο του 12ου Συνεδρίου της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Δικαστηρίων, τα συνταγματικά δικαστήρια είναι οργανωμένα σε ένα που συχνά διοργανώνουν συνδιασκέψεις, και πρόσφατα αφιερώσαμε τη συζήτησή μα στις σχέσεις μεταξύ των σωματικών δικαστηρίων και των υπόλοιπων δικαιοδοσιών, τόσο εθνικών όσο και διεθνών. Συγκεκριμένα τις σχέσεις μας με το δικαστήριο του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου. Αυτό είναι και ένα από τους λόγους που προσεκλήθην και με ιδιαίτερη τιμή συμμετάσχω στη σημερινή σας συζήτηση. Όπως ε, είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, το συγκεκριμένο ζήτημα που μας απασχολεί σε αυτό το μέρος της ακρόασης είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως θεσπίστηκε από τα ανώτατα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα αναφερθώ κυρίως στο Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου βεβαίως, αλλά θα σχολιάσω και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το Συνταγματικό Δικαστήριο βεβαιώνεται για την ε, τήρηση των υποχρεώσεων από τους διάφορους συνταγματικούς δικαστές του Βελγίου που είναι 7 με ίσο δικαίωμα ψήφου. Για την τήρηση λοιπόν των υποχρεώσεων σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως απαριθμώνται στο Σύνταγμα, στον τίτλο 2 και ορισμένα τα οποία ήδη έχουν ε, συμπεριληφθεί στο Σύνταγμά μας από το 1831. Το συνταγματικό δικαστήριο λοιπόν μπορεί να επιληφθεί μια υπόθεση με δύο τρόπου. Πρώτα απ' όλα, εφόσον υπάρξει προσφυγή επικυρώση μια συνταγματική πράξη μέσα σε προθεσμία έξι μηνών μετά την δημοσίευση τη νομοθετική πράξη στην επίσημη εφημερίδα. Η πρόσβαση είναι ευρεία είναι ανοιχτή στου προνομιούχου, όπω λέγονται, προσφεύγοντε, τι διάφορε κυβερνήσει δηλαδή, που μπορεί να υπάρχουν στο Βέλγιο, του προέδρους των κοινοβουλίων αλλά και τους ε, απλούς ενάγοντες, οποιοδήποτε φυσικό νομικό πρόσωπο δηλαδή, συμπεριλαμβανομένων των ε, ενώσεων, των μη κοινωνικοπικών οργανώσεων ή με δικαιολογημένο όφελος, που μπορούν δηλαδή να αποδείξουν ότι ενδεχομένως να πλήττονται εμέσως και δυσμενώς από τη διάταξη την οποία, κατά της οποίας προσφεύγουν. Η πρόσβαση λοιπόν είναι ευρεία για τα συνταγματικά δικαστήρια. Μπορεί επίσης κανείς να προσφύγει μέσω προδικαστικού ερωτήματος για οποιοδήποτε νομοθετική διάταξη, όποια και είναι η ημερομηνία της, συχνά μάλιστα Μας τίθενται ερωτήματα για την εφαρμογή του άρθρου 1382 του κώδικα αστικού δικαίου του 1804. Υπάρχει δηλαδή εκεί κάποιο θέμα με τη συνταγματικότητα ορισμένων κανόνων που προκύπτουν από αυτό το άρθρο. Τώρα, ο έλεγχος που ασκεί το δικαστήριο περιορίζεται στα δικαιώματα όπως αυτά, τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Σύνταγμά μας η απάντηση θα είναι μια απάντηση νορμανδού, διτή δηλαδή, και ναι και όχι. Σε ό,τι αφορά τα ουσιαστικά δικαιώματα, την ισότητα ως προς τα ποινικά ζητήματα, το σεβασμό του ιδιωτικού βίου και του οικογενειακού βίου. Για αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα τα ουσιαστικά δικαιώματα που συμπεριλαμβάνονται στο Σύνταγμα αλλά έχουν διάσταση ανάλογη, εμβέλεια ε, ανάλογη με τις πράξεις που προστατεύονται από διεθνή νομοθετήματα όπως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση το δικαστήριο θεωρεί ότι τα δικαιώματα αυτά εθνικής και διεθνούς εμβέλειας πρέπει να εξετάζονται από αυτή τη διτή προοπτική επειδή και στην εσωτερική μας νομοθεσία συνδέονται ιδιαίτερως με την ε, διεθνή εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτά. Αυτών. Και έτσι λαμβάνεται υπόψη και η νομοθεσία του δικαστηρίου του Στρασβούργου πολύ σοβαρά. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία. Πέραν των ουσιαστικών δικαιωμάτων στο Σύνταγμα, αναφέρεται ένα θεμελιώδης δικαιώμα που δεν θεωρείται ουσιαστικό, το οποίο κατά παραπομπή ορίζεται. Η ορχή η αρχή της νομιμότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Αρχή που πρέπει να τηρούν οι εθνικές νομοθεσίες ενώπιον κάθε άλλου δικαιώματος. Αστικές αρχές, ε, φορολογικές, δημοσίου δικαίου. Όμως, δεν μπορεί να υπάρξει διακριτική. Εάν μάλλον υπάρχει ζήτημα διακριτική μεταχείρισης, το δικαστήριο από το 1991 είπε ότι όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκύπτουν από διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει το Βέλγιο δεν μπορεί να υπάρξει εκεί διακριτική μεταχείριση που να προκύπτει από εθνική νομοθεσία. Συνήθω ε, οι περισσότερε αναδρομέ γίνονταν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και στο κοινοτικό κεκτημένο. Το δίκαιο δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπε και ο συνάδελφο, το δικαστήριο του Βελγίου ήταν το πρώτο συνταγματικό δικαστήριο που έθεσε προδικαστικό ερώτημα. που αφορούσε και την ερμηνεία και την εγκυρότητα δευτερογενού νομοθετήματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει πρωτογενέ δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτό προβλέπει το άρθρο 6 τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρώτη του παράγραφο κιόλα. Μπορούμε να πούμε ότι δεν αλλάζουν και πολύ τα πράγματα σε σχέση με το τι ίσχυε στο παρελθόν. Γιατί ήδη από το 1870 σε διεθνή απόφαση το δικαστήριο ορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν μέρος των γενικών αρχών όπου που προσφεύγουν οι δικαιοδοσίες για να εξασφαλίσουν την τήρηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κοινοτικές πράξεις. Η νομολογία αυτή εγκρίθηκε από τη συνθήκη του Μάστριχτ και η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παράγραφο 3 επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την τοποθέτηση. Αληθεύει βεβαίω ότι ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει την αρετή, παρουσιάζει την αρετή, να επιφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια παρουσιάζοντας έναν κατάλογο. Ακόμη και αν στο άρθρο 6 παράγραφος 3 ο κατάλογος αυτός δεν είναι διεξοδικός διότι θα μπορούσε να αναφέρεται και στι συνταγματικές παραδόσεις και στα διεθνή μέσα που διαθέτουμε. Ο τίτλος 7 της χάρτας με τίτλο «Γενικές διατάξεις σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή της χάρτας» είναι ίσως ο πλέον σημαντικός για τις εθνικές δικαιοδοσίες. Αντίθετα με ότι πίστεψαν κατά καιρού κάποιοι, ο χάρτης δεν προβλέπει ένα νέο σύστημα προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος να προστεθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Σύμφωνο αστική ε, Συνεργασίας και ούτω καθεξής. Όχι. Όλα τα εθνικά συντάγματα, κατά κανόνα, συμπεριλαμβάνουν μια παρήθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η χάρτα κάνει ακριβώς το ίδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι ομόσπονδο κράτος βεβαίως αλλά είναι μια ένωση κρατών. Είναι μια ένωση στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες για άσκηση δικαιοδοτικών καθηκόντων. Ο χάρτης λοιπόν προσφέρει ένα δυναμικό συνοδείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων επιβάλλεται στους εθνικούς νομοθέτες και στις κοινοτικές αρχές, στον κοινοτικό μάλλον νομοθέτη και τις κοινοτικές αρχές, αλλά και στα κράτη-μέλη όταν υλοποιούν το κοινοτικό δίκαιο. Το θύμισε ο συνάδελφος μόνον όταν υλοποιούν το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό επιβεβαιώνεται και στο άρθρο 51 της χάρτας. Η εθνική νομοθεσία και δεν θα σχολιάσω εδώ την εκτελεστική εξουσία πρέπει να σέβεται τις βασικές αρχές του χάρτη αλλά μόνον όταν υλοποιεί το δίκαιο της Ένωσης λόγου χάρη στην εκτέλεση κανονισμών ή στη μεταφορά οδηγιών. Για τους κανονισμούς σε σχέση με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για μη τήρηση του κανονισμού. Κάποιες φορές λέμε απλώς επιβάλλονται κυρώσει στα κράτη. Όμως οι κυρώσει αυτές πρέπει να σεβαστούν το συνταγματικό δίκαιο το εθνικό σε σχέση με, την, με το παράνομο και την προβλεψιμότητα των ε, παραβάσεων. Και το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και την παράγραφο 7 του αντίστοιχου άρθρου της Ευρωπαϊκής Χάρτας όπου λέγεται ότι οι κυρώσεις δεν μπορεί να είναι δυσανάλογες σε σχέση με τη σοβαρότητα της παράβασης. Όμως οι διατάξεις αυτές τόσο ή καλύπτονται από την ομολογία του Στρασβούργου. Σε ό,τι αφορά τις οδηγίες έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε την υλοποίηση του στόχου αλλά έχουμε στην νομοθεσία μεταφοράς νησοδηγίας και ένα περιθώριο ελιγμών. Το οποίο αφήνει στα κράτη-μέλη ενίοτε κάποιες ελευθερίες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω δεν εφαρμόζεται η χάρτα, αλλά το συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών. Το άρθρο 52 είναι εξαιρετικά σημαντικό για το εύρος και την ερμηνεία των δικαιωμάτων και αρχών. Στην παράγραφο 2 και 3 ιδιαιτέρως. Στο βαθμό όπου ο χάρτης συμπεριλαμβάνει δικαιώματα που ανακαλύπτονται και από την σύμβαση, η ουσία τους συμπίπτει με αυτήν που τους προσδίδει η σύμβαση. Κατά κυριολεξία, η αρχή αυτή είναι πολύ όμορφη, αλλά δεν είναι πολύ σαφής. Διότι ποια είναι ακριβώς η εμβέλεια της σύμβασης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν καταλαβαίνουμε την εμβέλεια της σύμβασης αναγυγνώσοντας κάποια από τα άρθρα της σύμβασης, αλλά μόνον εάν μελετήσουμε την ομολογία του Στρασβούργου. Νομίζω λοιπόν ότι για να αποτιμήσει κανείς την εγκυρότητα του εθνικού δικαίου κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου, το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να μεταφέρει την νομολογία εάν χρειαστεί και να μην θέτει προδικαστικά ερωτήματα στο Λουξεμβούργο. όταν το εθνικό δίκαιο πρέπει να σεβαστεί ταυτόχρονα μια διάταξη της χάρτας και μία της σύμβασης που αφορούν το ίδιο θέμα. Αλλά ακριβώς ε, αυτό καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο του Στρασβούργου και εάν χρειαστεί μπορεί να αναδράμει κανείς αυτήν την διάταξη. Δεν θα περάσω και στο δευτερογενέ δίκαιο εδώ, αλλά σε κάποιε απορίες. Ο χάρτης απαριθμεί δικαιώματα και ελευθερίες, τα οποία θεωρούνται τεκμηριωμένα και επίσης κάποιες αρχές σε θέματα οικονομικά και κοινωνικά, όπως τον οποίων μάλλον το εύλογο είναι κάπως περιορισμένο. Εδώ με την ε, απλή ανάγνωση της, ε, τουλάχιστον του χάρτη δεν μπορεί κανείς να καταλήξει στις δύο κατηγορίες διατάξεων που περιλαμβάνει τόσο εύκολα. Η έλευση του χάρτη ίσως οδηγήσει τις εθνικές δικαιοδοσίες να θέσουν νέα προδικαστικά ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα για το δικαστήριο αυτό θα είναι σε θέση να ε, ανταποκριθεί σε τέτοια συρροή ερωτημάτων. Διότι αν δεν αποφασίσουν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα οι δικαιοδοσίε εθνικέ, ε, το ορίζει στο άρθρο 47 η σύμβαση, τότε μπορούν να τρέξουν σε προδικαστικό ερώτημα. Μεταξύ 18 και 24 μηνών πρέπει να απαντήσει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της χάρτας και της σύμβασης να πω ότι σε αντίθεση με όσα κατά καιρούς δηλώθηκαν το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο δεν είναι ισότιμα. Το Λουξεμβούργο εξασφαλίζει τα θεμελίδια δικαιώματα σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο και το Στρασβούργο σε σχέση με το εθνικό. Όχι όμω, Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα όργανο δικαστικό, δικαιοδοτικό, το ανώτατο που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομική οντότητα και με τις αρμοδιότητες που τις έχουν εκχωρήσει τα κάτι μελη ενώ το δικαστήριο του Στρασβουργού επαγρυπνεί για όλες τις δραστηριότητες των κατομελών Είτε ασκούνται σε επίπεδο εθνικό είτε συλλογικά. Και αυτό και πριν την προσχώρηση, όπως είπε ο συνάδελφος από το δικαστήριο, από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Το γεγονός ότι εκτελείται το κοινοτικό δίκαιο δεν μας απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δικαστήριο του Στρασβούργου, βέβαια με να μην φανταστεί ότι ήθελα να του υποκαταστήσω, εάν δεν βρίσκονταν εδώ, απλώς ήθελα να σχολιάσω κι εγώ ένα μέρος του ρόλου τους. Παρουσία του Πρόεδρου Κώστα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μελκιόρ. Και τώρα, η τελευταία παρέμβαση για αυτό το μέρος της Συναντησή μα από τον κύριο Μάρκ Μποσουή, πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Βελγίου, επιτετραμένου για τα θέματα προσφύγων και ασύλου. Πρόεδρε, έχω ετοιμάσει την ομιλία μου στα γαλλικά. Σε ό,τι αφορά τι σχέσει με τις ανώτατες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες, το Βελγικό Συνταγματικό Δικαστήριο τηρεί μια στάση πλήρου συνεργασία εξετάζοντας το κατά πόσον η βελγική νόμη είναι συμβατή με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που εξασφαλίζει το Σύνταγμα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου έχει, παρα, έχει διευρύνει τον ελεγχό του εξετάζοντας τις νομοθετικές διατάξεις σε σχέση με δικαιώματα και ελευθερίες που είναι ανάλογες και διασφαλίζονται από διεθνείς συμβάσεις όπου έχει προσχωρήσει το Βέλγιο. Για το σκοπό αυτό έχει συμπεριλάβει και την ίδια την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ό,τι αφορά το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνταγματικό δικαστήριο απευθύνεται στο δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όποτε ανακύπτει ένα θέμα νομιμότητα ή ερμηνεία δικαιώματο που έχει σχέση με το δικαίωμα μάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου έχει θέσει 10 προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο του Λουξεμβουργού, έναν αριθμό ανώτερο από το σύνολο των υπόλοιπων συνταγματικών δικαστηρίων όλων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί. Αυτή η συμπεριφορά μόνιμης συνεργασίας δεν εμποδίζει βέβαια να ανακύπτουν απορίες σε σχέση με κάποιες από τις πρόσφατες εξελίξεις και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες. Σε ό,τι αφορά το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, στη χώρα μας, όπως και σε άλλα συνταγματικά δικαστήρια, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που έχουν να κάνουν με την χρήση που ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε ο χάρτης των, θεμελιδών δικαιωμάτων της Ένωσης με την αφορμή πρόσφατων προδικαστικών ερωτημάτων που έχουν θέσει οι βελγικές και γαλλικές εθνικές δικαιοδοσίες, είναι σημαντικό να θυμίσουμε, όπως και ο πρόεδρος ε, Μελχιόρ έκανε ήδη, ότι ο χάρτης αφορά τα θεσμικά όργανα τα, και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας και στα κράτη-μέλη, αλλά μόνον κατά την υλοποίηση του δικαίου της Ένωσης δεν θα άρμοζε το δικαστήριο του Λουξεμβούργου βασιζόμενο στο χάρτη αυτό να εξετάζει τα ερωτήματα που έχουν θέσει οι εθνικοί δικαστές ό,τι αφορά τους κανόνες του εσωτερικού δικαίου εφόσον δεν αφορούν την υλοποίηση του δικαίου της Ένωσης αλλά που θα θεωρούνταν από τους εθνικούς δικαστές ενδεχομένως ως αντικείμενοι στα αντίθετη μάλλον με τα δικαιώματα του ανθρώπου όπως θα διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Αυτό θα μπορούσε να πλήξει τις ε, αρμοδιότητες και των συνταγματικών δικαστηρίων από τη μία και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την άλλη. Σε προσωπικό τώρα επίπεδο θα ήθελα να τονίσω ότι είμαι ένθερμος οπαδός, ε, ανέκαθεν μάλιστα, της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μου φαίνεται παρόλα αυτά συνετό να ε, συμμετάσχουν όλα τα, να είχαν συμμετάσχει όλα τα συνταγματικά δικαστήρια των εθνικών κρατών μελών στις σχετικές συζητήσεις και για τη διαδικασία προσχώρησης προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ρόλοι και αρμοδιότητες των ΜΕΝ και των ΔΕ σε σχέση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά το δικαστήριο του Στρασβουργού, νομίζω ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει το δικαστήριο αυτό λόγω του πολύ αυξημένου αριθμού, πάνω από 125.000, και αριθμού που συνεχώ αυξάνεται των υποθέσεων που ακόμη δεν έχουν εκδικαστεί. Προσωπικά, πρόσφατα δημοσίευσα ένα άρθρο στην Human Rights Law Journal για την ε, διεύρυνση μέσω της εκτελεστικής εξουσίας, της δικαιοδοσίας ε, του Δικαστηρίου των ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων και από την άλλη ενός βιβλίου στις εκδόσεις Brillant με τον τίτλο οι δικαστέ σε όλη τη οδόστρωμα σε σχέση με τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου ό,τι αφορά το θέματα ασύλου και του ετούντε άσυλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον διπλά επικουρικό χαρακτήρα τη δικαιοδοσία των ευρωπαϊκών δικαιοδοσιών, από τη μια πρέπει να σκεφτούμε ότι τι αρμοδιότητε αυτέ ασκεί ο εθνικό νομοθέτη και από την άλλη οι εθνικέ δικαιοδοσίε. Ε, εγώ ήμουν ε, υπέρ του να ε, επιδείξουμε περισσότερη σύνεση και επιμέλεια, καθώς και εγκράτεια και επιφυλακτικότητα. Αναγνωρίζοντας ότι η σύμβαση πρέπει να ερμηνεύεται υπό το φως του ισχύοντος πλαισίου, και ότι δεν σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει θεωρητικά δικαιώματα ή απατηλά δικαιώματα, αλλά δικαιώματα πρακτικά και χειροπιαστά, μου φαίνεται σε αυτή την περίπτωση ότι το να διευρυνθεί η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και στον τομέα τη κοινωνική ασφάλεια, ε, υιοθετώντα μια ερμηνεία πολύ ευρεία του δικαιώματο ε, ιδιοκτησία, αυτό θα καταργούσε κάθε περιορισμό στι αρμοδιότητε του δικαστηρίου πέραν των περιορισμών που το ίδιο το δικαστήριο θέτει στον εαυτό του. Όπως δει το δικαστήριο δρά και ως διεθνής δικαστής, ελέγχοντας τη συμβατότητα με τις διατάξεις της σύμβασης, καθώς και με την νομοθεσία των κρατών που συμμετέχουν, σε σχέση με την ε, νομολογία των ανώτατων κρατικών δικαστηρίων. Όμως κάποιες φορές ε, το δικαστήριο ενεργεί και ως δικαστής έφεσης όταν το απαιτεί η υπόθεση ή και ε, δικαστής ακύρωσης ε, ξεκριβώνοντας αν έχει εφαρμοστεί σωστά το εσωτερικό δίκαιο ή και όπως από το 2004 έχει συμβεί και ως δικαστής για ασφαλιστικά μέτρα επιβάλλοντας τέτοια δεσμευτικά ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν <clears throat> είναι μια καινοτομία ότι τα, οι αιτήσει εκθέσεις του δικαστηρίου έχουν επιφέρει μια σοβαρότατη αύξηση των αιτήσεων για την υλοποίηση των προσωρινών μέτρων. Από το 2008 περίπου 3.200 τέτοιες αιτήσει υποβλήθηκαν και το δικαστήριο το ίδιο μας έχει πει ότι συνήθως αυτό αφορά ευαίσθητες υποθέσεις που έχουν να κάνουν τα δικαιώματα των αλλοδαπών και των ετούντων άσυλο και πολλές φορές απαιτούν πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να εξεταστούν τάχιστα. Τα προβλήματα του δικαστηρίου μπορεί να επιδεινωθούν εάν πολλά κράτη-μέλη κυρώσουν το 12ο πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης διότι εκεί περιέχεται μια γενική απαγόρευση τη διακριτική μεταχείριση. Προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα τη ατομική προσφυγή, ένα από, τα, ένας από τους ακρογωνιαίους λήθους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα έπρεπε νομίζω σε αυτή την περίπτωση να έχουμε μια πολύ σοβαρή μελέτη του θέματος αυτού στο πνεύμα της συνδιάσκεψης του Ιντερλάκεν για το ρόλο ακριβώς του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και για το ποιος, πώς θα πρέπει να εξελιχθεί αυτός ο ρόλος στο μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, uh, Σας ευχαριστούμε. Είχαμε τρεις ε, παρεμβάσεις, τρεις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις όσον αφορά τον ρόλο και τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του ΔΕΚ στο Λουξεμβούργο και τον συσχετισμό του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και του ΔΕΚ στο Λουξεμβούργο. Και όταν εδραζόμαστε και επικεντρωνόμαστε τώρα σε σχέση με τη συζήτηση σε αυτά τα θέματα, θα ήθελα να ζητήσω πρώτα από τον συνάδελφο που θα ήθελε να παρέμβει, τον κύριο Τόντο που ήταν εισηγητής εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σε σχέση με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τους προβληματισμούς και τις σκέψεις που παρουσιάστηκαν από πλευρά των εισηγητών και σίγουρα πρέπει να πω ότι έχουν επιπτώσεις σε σχέση με θέματα τα οποία είχαν, στα οποία είχαν επικεντρωθεί οι συζητήσεις μας και σε σχέση και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και εμείς στη Συνταγματική, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είχαμε επικεντρωθεί σε αυτά τα θέματα όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζετε αυτή η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες και σίγουρα πτυχές όπως αυτές που παρουσιάσατε και θέσατε εσείς θα είναι αντικείμενο συζήτησης μέσα σε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Εγώ ιδιαίτερα έχω κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να σας διατυπώσω διότι ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλές αμφιβολίες για αυτά τα θέματα που είναι τόσο σημαντικά. Από την άλλη πλευρά όπως η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση αυτή και στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Η πρώτη ερώτηση που ήθελα να διατυπώσω είναι ακριβώς αν εσείς θεωρείτε ότι θα είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια προηγούμενη οδός ε, πρόσβασης ή προσφυγής ε, στο 10 του Λουξεμβούργου στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν θα έχουν εξαντληθεί δυνατότητες προσφυγές μέσω των εθνικών δικαστηρίων που θα μπορούσαν να παρέμβουν. Όταν υπάρχει εδώ αμφισβήτηση ή θέμα μιας κοινοτικής πράξης και έχει εξαντληθεί η διαδικασία στα εθνικά δικαστήρια, τι θα μπορούσε να γίνει μετά. Διότι όπως ακριβώς προβλέπεται από τις διατάξεις μας, προβλέψιμο είναι ότι αν ένας πολίτης, ας υποθέσουμε Γερμανός, αμφισβητήσει μια ευρωπαϊκή πράξη, μια διάταξη ευρωπαϊκή όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξαντλήσει όσον αφορά το συνταγματικό δικαστήριο της Καλσρούης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας τις δυνατότητες προσφυγής θα μπορούσε να περάσει άμεσα στο 10 <clears throat> ώστε εκεί να μπορέσει να τύχει συνέχεια η προσφυγή. Αλλά αυτό τι θα σήμαινε σε σχέση με το δικαστήριο το 10. Και σε αυτό πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα το οποίο τίθεται. Διότι θεωρητικά δεν θα ήταν λογικό λόγω ε, αμφισβήτησης ε, όσον αφορά την, ε, τις αρχές ε, της σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κανείς να μην μπορεί να προσφύγει στο ΔΕΚ χωρίς να έχει προηγούμενα προσφύγει στο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Πραγματικά θα έπρεπε να θεσπιστεί αυτή η προηγούμενη απέτηση. Το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο πρόβλημα της διασύνδεσης μεταξύ χάρτας και σύμβασης. Διότι όπως πολύ καλά είπατε εσείς ε, ως προλαλή σας, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη ως προβληματισμός για το ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία εμπεριέχει η χάρτα που δεν είναι τόσο ρητά, δεν αναφέρονται τόσο ρητά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η χάρτα μετατρέπεται σε κοινοτικό δίκαιο, σε πρωτογενές δίκαιο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει σε μια σύμβαση, όμως όχι σε όλα τα πρωτόκολλα αυτής της ε, σύμβασης. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω είναι ποια από τα πρωτόκολλα αυτά που συμπληρώνουν, ολοκληρώνουν την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή αυτή σύμβαση και που εξελίχθηκαν κατά, τη διάρκεια των ετών, θα έπρεπε να αναπτυχθούν υποχρεωτικά στην προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση. Ποια θα εμπεριέχονται σε αυτή, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί απλά να διαπραγματευτεί την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όχι όμως σε όλα τα πρωτόκολλα. Η ερώτηση, ποια τα πρωτόκολλα αυτά είναι υποχρεωτικά, υποχρεωτικής εφαρμογής όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει συνεκτικότητα και συνάφεια με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η τρίτη ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω. Με ποιο τρόπο ακριβώς επιλύεται η αντίφαση στην προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πρωτόκολλα της Σύμβασης ώστε να μην αλλοιώνεται η ουδετερότητα εκείνων των χωρών που δεν έχουν προσυπογράψει τη χάρτα. Διότι εδώ υπάρχει η αρχή opting out, αυτοεξαίρεσης όσον αφορά ε, τη χάρτα ε, αυτή. Οι τρεις χώρες που όπως γνωρίζετε δεν έχουν προσυπογράψει και στις οποίες δεν εφαρμόζεται η χάρτα αυτή. Με ποιο τρόπο λοιπόν η αρχή του πρωτοκόλου που θεσπίζει ότι η προσχώρηση δεν θα αλλοιώνει την ουδετερότητα ως χαρακτηριστικό των χωρών της Ένωσης. Τι θα γίνει με αυτό. Θα περιοριστεί η δυνατότητα η διαπραγματευτική της ε, ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τέλος η τέταρτη τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω είναι η έξοεδαφική εφαρμογή της ε, ευρωπαϊκής αυτής σύμβασης. Και αυτό διότι όταν θα προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την σύμβαση θα το κάνει υπό το πρίσμα της δράσης και δραστηριοποίησής της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Α υποθέσουμε οι στρατιωτικέ δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνεί δράσει και πρωτοβουλίε ή ας υποθέσουμε ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την ανάπτυξη, τι πρεσβείε, την εξωτερική υπηρεσία, διπλωματική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αρχίσει να λειτουργεί τώρα και τέτοιε περιπτώσει. Θεωρώ ότι η έξω εδαφική εφαρμογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους, ε, τα θεσμικά τη όργανα υπάρχει ω υποχρεωτικό χαρακτήρα τη υλοποίηση των αρχών αυτών της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και για τις αρχές της σύμβασης αυτής και των πρωτοκόλων της. Με ποιο λοιπόν τρόπο θα μπορεί να απαιτεί κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμογή, την υλοποίηση αυτών των αρχών και Ποιο και πότε θα γίνεται αυτό. Όταν για παράδειγμα ένας βολιβιανός πολίτης ε, θα διεκδικεί και θα πηγαίνει στο δικαστήριο του Στρασβούργου για τη δράση ενός όργανου ανάπτυξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση στη Βολιβία που όταν αυτός ο Βολιβιάνος ή αυτοί οι Βολιβιανοί θα θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ή έχουν παραβιαστεί αρχέ τη χάρτα, ε, παράδειγμα για μια κοινότητα ηθαγενών κτλ αυτή η εφαρμογή εξοεδαφική θα ήθελα να μου την αναπτύξετε περισσότερο σένια. Αυτά είχα να πω Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις εισηγήσεις σας κύριε. Thank uh, ε, Έχουμε τώρα όλες αυτές τις ερώτησεις ε, που διατυπώθηκαν και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι περίπλοκο το θέμα της ε, συνεδρίασής μας και μετά την δυνατότητα που θα υπάρξει να απαντηθούν αυτά τα θέματα και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα τεθούν αυτά τα θέματα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν τώρα. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους εισηγητές και μετά να προχωρήσουμε για περαιτέρω ερωτήσεις ε, και παρεμβάσεις από τα μέλη τους παρόντες στην αίθουσα. Πρώτα λοιπόν ο κύριος Μποσό και ο κύριος Μελκιόρ και ο κύριος Μωσή. Προσπαθήστε αν θέλετε να απαντήσετε τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Αν μπορείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως λέμε στη γλώσσα μου, όταν κάτι είναι δύσκολο και δύσκολο μπορεί να απαντηθεί, λέει κάποιος «Α, εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που ρωτήσατε». Είναι ε, καταλητική σημασία στο ερώτημά σας για την ε, ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δώσω μία απάντηση, συνοψίζοντας, θα έλεγα πως δεν πρέπει να προσπαθούμε να οργανώσουμε την αταξία. Τι σημαίνει αυτό. Απαραίτητα πρέπει να βρούμε τα μέσα εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας που είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμογή αυτής της αρχής με τον ίδιο τρόπο ή τουλάχιστον με όχι λιγότερο αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με την εφαρμογή του στα κράτη-μέλη. Δηλαδή να ισχύει η αρχή της αλογικότητας με τον ίδιο τρόπο για την Ένωση και για τα κράτη-μέλη. Για να διευρύνω τον προβληματισμό θα έλεγα ότι αρμόζει στη συμφωνία προσχώρησης να έχουμε σαφείς κανόνες. Φερρυπίν, όταν έχει τεθεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πρέπει να περιμένουμε την απάντηση του δικαστηρίου και να περιμένουμε ε, ο εθνικός δικαστής ε, να λάβει υπόψη με τη δική του απόφαση αυτήν την σύμβουλη της, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πρέπει να καλύψουμε την περίπτωση όπου δεν θα έχει τεθεί ένα προδικαστικό ερώτημα. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Κάτι άλλο και εδώ επιμένω. Θα ήταν θεμητό για μια εθνική δικαιοδοτική αρχή να λάβει υπόψη την ομάδα των, ε, που σχετίζεται με τα προδικαστικά ερωτήματα τα τελευταία 50 χρόνια. Δηλαδή μια εθνική δικαιοδοτική αρχή στα πλαίσια της απόφασης Ιλφίτε που, ε, από την 6η Οκτωβρίου 82 μπορεί να αποφασίσει εν πάση περιπτώσει μια εθνική δικαιοδοτική αρχή να μην υποβάλει ε, προδικαστικό ερώτημα. Ωραία, εν τη αυτή περιπτώσει χρειάζεται ένας μηχανισμός ώστε όταν δεν καλείται να αποβαθανθεί το δικαστήριο, παρόλα αυτά να έχετε δυνατότητα να εκπληρώσει την αποστολή του. Παραδείγματο χάρη, ακούστηκε η ιδέα, αλλά βέβαια δεν είναι και η μόνη λύση, πρέπει να σκεφτούμε και άλλε πιθανέ λύσει. Ακούστηκε λοιπόν η εξή ιδέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι ενώπιον του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Δηλαδή, να πει ας αφήσουμε να αποφανθεί το δικαστήριο του Λουξεμβούργου και αν ε, κάποιος διάδοκος δεν είναι ικανοποιημένος με την έκβαση της απόφασης, τότε μπορεί να αποταθεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό μπορεί να διευρυνθεί ε, και στα κράτη-μέλη. οι διάδικοι ενώπιον του Εθνικού Δικαστή μπορεί να επικαλεστούν το δικαίωμα εξαίρεσης από τον ενωσιακό έλεγχο. Αυτό που πρέπει να ε, κατοχυρώσουμε είναι ότι όλοι θα μπορούν να εκπληρώνουν την αποστολή τους. Είπαμε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχει την νομιμότητα των νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Το δικαστήριο του Στρασβούργου δε καλείται να αποφανθεί κατά την εφαρμογή αυτών των νομοθετημάτων για ενδεχόμενες παραβιάσεις ε, των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι εξαιρετικά περίπλοκα και τεχνικά αυτά τα ζητήματα και ορισμένες φορές αποφεύγουμε να ε, καταπιαστούμε με κάποια ζητήματα. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε το ζήτημα της εγκυρότητας, της νομιμότητας ε, των ε, νομοθετημάτων ε, θα πρέπει να εξεταστεί από κοινού με το θέμα της ερμηνείας. Διότι η ερμηνεία που δίδεται από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου μπορεί να οδηγήσει στη διαπίστωση ότι είναι παράτυπη μια νομοθετική πράξη Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εφαρμογή της. Είπε ο συνάδελφος ότι το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας του έκανε, έστειλε συρροή ε, προδικαστικών ερωτημάτων. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν και άλλα τέτοια προδικαστικά ερωτήματα, όπως για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, ε, προδικαστικό ερώτημα που προέρχεται από τη Γαλλία. Το δικαστήριο ερμηνεύει μέσα από αυτά τα προδικαστικά ερωτήματα τις διάφορες οδηγίες ε, και μάλιστα είπε τα δικαστήρια σε μια συγκεκριμένη υπόθεση ότι δεν μπορούμε να θεσπίζουμε υποχρέωση καταγγελίας από πλευρά ενός ε, δικηγόρου όταν ο δικηγόρος ε, αποτιμά την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πελάτης ή όταν υπερασπίζεται τον πελάτη ενώπιον μιας εθνικής δικαιοδοτικής αρχής δεν μπορεί να υποχρεωθεί να τον καταγγείλει ταυτόχρονα. Προκαταλήψεις δεν έχουμε πάντως. Το μόνο που ισχυριζόμαστε και το μόνο που θέλουμε να υποδείξουμε και στον Ευρωπαίο νομοθέτη και σε όσοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο αυτών των ζητημάτων είναι ε, να βρούμε λύσεις και αυτές οι λύσεις θα περάσουν μέσα από τους κανόνες της Συμφωνίας Προσχώρησης στην ε, Σύμβαση ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόεδρε, θα θέλατε να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα. Μάλιστα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Για το δεύτερο ερώτημα του πεδίου εφαρμογή, μα όπως και τα άλλα, είναι πολιτικό ζήτημα. Έκανα ε, μία ε, μελέτη για τη σχέση ανάμεσα στη σύμβαση και τα πρωτοκολλά της αφενός και της χάρτας αφετέρου. Λοιπόν, ε, και κατέληξα στο εξή συμπέρασμα. Αν ε, συνδυάσουμε τη σύμβαση με τα πρωτόκολλα, κατά 80% περίπου καλύπτουμε την ε, χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά είναι και θέμα επιλογή έτσι των πρωτοκόλλων στα οποία θα προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου και μια παρένθεση. Είπαν οι συνάδελφοι πολύ σωστά ότι η χάρτα εμπεριέχει ε, διατάξεις που υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Λέμε ότι δεν πρέπει να επιβάλλουμε τη θανατική ποινή. Ευτυχώ, ευτυχώ, προς το παρόν, τα θεσμικά όργανα τέτοια εξουσία, τέτοια αρμοδιότητα δεν έχουν ε, στον τομέα του ποινικού δικαίου. Δεν μπορούν να επιβάλλουν ε, την ανώτατη ποινή. Τέλο πάντων είναι ε, πολιτική απόφαση. Το ίδιο ισχύει, αν και είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα, το ίδιο ισχύει λοιπόν και για κάποια κράτη και το πώς τοποθετούνται σε σχέση με την ε, χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να δούμε αυτά τα κράτη. Πώς, ποια σχέση έχουν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει μια σχετική μελέτη. Εγώ δεν ασχολήθηκα με το ζήτημα προς το παρόν. Εξάλλου υπάρχουν και άλλοι αρμοδιότεροι που θα μπορούσαν να ε, μελετήσουν αυτό το θέμα της εμβέλειας ε, της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Για την εξοεδαφικότητα τώρα, να σας δώσω μία πρώτη κατά προσέγγιση απάντηση. Η χάρτα σχετίζεται με θεσμικά όργανα που δεσμεύονται μέσα από τη σύμβαση, όποιος και αν είναι που καταγγέλει αυτή την παραβίαση των δικαιωμάτων του. Στην ομολογία του ε, δικαστηρίου, για να, πρέπει οπωσδήποτε μάλλον, ε, εννοεί ο μιλητή, να λάβουμε υπόψη την ομολογία του δικαστηρίου για να ερμηνεύσουμε σωστά τις σχετικές διατάξεις. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Μελκιόρ, μήπως ε, θα θέλετε κι εσείς να παρέμετε και να δώσετε ενδεχομένω κάποιες ε, απαντήσεις. Ευχαριστώ. Όταν μια κοινοτική πράξη καταγγέλλεται στο Στρασβούργο επί παραβάση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ερώτημα είναι θα πρέπει να υπάρξει πρώτερη παρέμβαση η προσφυγή στο Λουξεμβούργο. Νομίζω, εάν η κοινοτική πράξη θεωρείται εκτός νόμου, εάν θεωρεί μια δικαιοδοσία ότι είναι εκτός νόμου, η εθνική δικαιοδοσία δεν μπορεί να αποφανθεί μόνη. Πρέπει να υπάρξει προδικαστικό ερώτημα που να έχει τεθεί στο Λουξεμβούργο και το Λουξεμβούργο μπορεί να πει ότι όχι, η πράξη αυτή σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όμω θα έχει όντω παρέμβει προηγουμένω στο Λουξεμβούργο. Τίποτα δεν εμποδίζει ωστόσο ο δικαστής του Στρασβουργού και σε σχέση με το σεβασμό του ίδιου θεμελιώδους δικαιώματο από την ίδια πράξη να έχει διαφορετική ερμηνεία. Δεν θα έχει τίποτα το περίεργο κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα προκύπτει όταν η κοινοτική πράξη σε εσωτερικό επίπεδο και εάν χρειαστεί έχει χαρακτηριστεί από το Εθνικό Δικαστήριο χωρίς να τεθεί προδικαστικό ερώτημα και τότε παραπέμπεται στο Στρασβούργο. Η νομιμότητα της κατάστασης δεν είναι πάντοτε προφανής λοιπόν. Θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα στο πρωτόκολλο να προβλέπετε κάποια δυνατότητα προδικαστικού ερωτήματος για παρέμβαση. της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ιδίας βάσει της διαδικασίας του Στρασβούργου. Μεταξύ χάρτας και σύμβασης τώρα. Ποια είναι τα πρωτόκολλα που πρέπει να συμπεριληφθούν. Υπάρχουν δύο είδων πρωτόκολλα. Τα συνταγματικά που τροποποιούν τη λειτουργία της σύμβασης και προφανώς πρέπει να εγκριθούν, να κυρωθούν αυτά και τα ουσιαστικά πρωτόκολλα. Εκεί κάνουν κάποια επιλογή τα κράτη-μέλη. Κάποια δεσμεύονται από πολλά, το Βέλγιο λόγω χάρη δεν δεσμεύεται ακόμα από το 7ο πρωτόκολλο, που είναι αρκετά παλιό παρόλα αυτά. Αλλά δεν προκαλεί πλέον προβλήματα στο Βέλγιο. Αλλά αυτό είναι και θέμα επιλογής. Το πρώτο πρωτόκολλο θα έλεγα ότι αξίζει τον κόπο. Διότι εκείνος το 1950 δεν είχε σωματωθεί γιατί προκαλούσε σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Και το πρόσθετο αυτό πρώτο πρωτόκολλο όπως ονομάζεται, αν και υπήρξαν και άλλα, Ονομάζεται απλώ πρόσθετο πρωτόκολλο, αλλά υπήρξαν το μεταξύ και άλλα, γι' αυτό πήρα τη σειρά του πρώτου. Ε, ε, ε, τώρα πια μπορεί να συμπεριληφθεί. Τώρα, χώρε που βρίσκονται σε ιδιαίτερη θέση λόγω τη προσχώρηση. Έναντι τη χάρτα, ναι, αλλά δεσμεύονται και από το άρθρο 6 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ούτω ή άλλω είναι συμβαλόμενα μέρη τη σύμβαση, τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν βλέπω λοιπόν τι έχει να φοβηθεί κανεί. Και ω προ την εξωτερική εφαρμογή, εκτό Ένωση, εδώ η δικαιοδοσία του Στρασβούργου δεν είχε πολλέ τέτοιε περιπτώσει να εξετάσει. Και δεν θα τοποθετηθώ επί της νομολογίας. Ευχαριστούμε κύριε Μπόσουιτ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα απαντήσω στα Ολλανδικά. Αλλά θα χρειαζόμουν μια γαλλική πρόταση επιπλέον. Θα ήθελα να αναφέρω να αναφερθώ στο αυτό το οποίο είπε ο προλαλής σας. Δεν πρέπει να οργανώσουμε, διοργανώσουμε το χάος. Μπορούμε νομίζω να συμφωνήσουμε όλοι επί, επαφής αυτής της Ένα πράγμα είναι σημαντικό. Το άρθρο 51 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με αυστηρό τρόπο ερμηνεύεται. Έχουμε την λέξη uniquement, μόνο ή αποκλειστικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αν δεν το προσέξουμε αυτό μπορεί πραγματικά το αποτέλεσμα να είναι μια χαοτική, χαόδης κατάσταση. Υπάρχει και ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο. Έχουμε τη σειρά, την αλληλουχία των διαφορετικών μέτρων ή βημάτων. Ένα παράδειγμα αναφέρθηκε. Επρόκειτο για το θέμα του μετά από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της ε, Συνταγματικό Δικαστήριο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας θα πρέπει να πάμε στο Στρασβούργο ή στο Λουξεμβούργο. Καλό θα ήταν από την Καρσρούη να μπορούσαμε να μεταβούμε στο Λουξεμβούργο. Είναι ακαθόδες όμως το θέμα αυτό. Πρέπει πρώτα το θέμα αυτό να διατυπωθεί, το ζήτημα αυτό να διατυπωθεί προς το Λουξεμβούργο, στο 10 όταν πρόκειται για θέμα ε, ερμηνείας ακριβώς. Και για το δεύτερο θέμα ήταν το θέμα για τα πρόσθετα πρωτόκολλα ε, υποδεσμευτικό χαρακτήρα. Έχουμε τα ρυθμιστικά πρωτόκολλα και σίγουρα δεν είναι πρόδειλο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσυπογράψει και να προσχωρήσει σε πρωτόκολλα στα οποία δεν μπορούν να ενταθούν και να προσυπογράψουν αυτά όλα τα κράτη-μέλη. Το θέμα των πρωτοκόλων λοιπόν με αυτή τη διαφοροποίηση πρέπει να απαντηθεί. Τώρα, για τις ε, χώρες που έχουν ένα, μια αυτοεξαίρεση, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό ως εξής. Δεν μπορεί κανείς να στραφεί στο Λουξεμβούργο στο 10 αν υπάρξουν προβλήματα τα οποία θα αφορούν τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θα είναι δυνατόν λοιπόν να θέσουν ένα τέτοιο ερώτημα, ένα τέτοιο αίτημα προς το Λουξεμβούργο. Θα πρέπει άμεσα να περάσουν προς το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, χωρίς εμπλοκή του ΔΕΚ στο Λουξεμβούργο. Και το θέμα της ε, εξοεδαφικής ε, ε, εφαρμογής και όσον αφορά την δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις ε, ε, μιας τέτοιας εξοεδαφικής εφαρμογής όσον αφορά τα κράτη-μέλη και αυτό αφορά τα ίδια τα κράτη-μέλη όπου έχουν υπογράψει αυτή την σύμβαση. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις παρεμβάσεις. Ο κύριος Κλέης. Σας ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω λόγο για τη διαφοροποίηση της δικαστικής δικαιοδοσίας, δικαστικής εξουσίας και όσον αφορά την, το νομοθετικό, την νομοθετική συνιστόσα αφενός και την, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφετέρου. Είναι δυσδιάκριτες οι διαχωριστικές γραμμές και απορρέουν προβλήματα για εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν αυστηρότερους ε, ε, κανονισμούς και διατάξεις όσον αφορά την πολιτική για τη μετανάστευση π.χ. για ελάχιστους ε, μισθούς ε, για ε, τέτοιους εργαζόμενους ε, μετανάστες που για παράδειγμα κάποιοι από αυτούς έχουν παντρευτεί υπήκο Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι σε σχέση με την ίδια τη μετανάστευση και τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών υπάρχουν επιπτώσεις και σε σχέση με τα κοινωνικά συστήματα ασφάλισης. Υπάρχει ζήτημα και διαφύλαξης, διασφάλισης των συστήματων αυτών. Πρόκειται όμως για δημοκρατικά αποφασισμένα μέτρα τα οποία ισχύουν με αυτόν τον τρόπο σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο. Αυτά τα μέτρα όμως, ας το πω έτσι, απαλήφονται λόγω της νομολογίας ε, στο, του δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο ή λόγω τη νομολογία του 10 στο Λουξεμβούργο. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, όμω κάτι τέτοιο είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη όταν όλα αυτά εξαλείφονται. Διότι είναι κυρίαρχε δημοκρατικέ αποφάσει κρατών μελών που έχουν θεσπίσει τέτοιου είδου αυστηρέ διατάξει. Όταν σε ένα υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτέ καταστρέφονται, υπονομεύονται, έρονται μέσω δικαστικών αποφάσεων, μέσω νομολογία, ε, τότε τίθεται το θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών, τα οποία υπονομεύονται στα εν λόγω αυτά θέματα. Και υπάρχει πρόβλημα εδώ και όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις ε, αυτών των αποφάσεων για αυτά τα κράτη-μέλη. Και έτσι βλέπουμε ότι η δικαστική δικαιοδοσία άμεσα έχει επιπτώσεις ε, στα κράτη-μέλη. Και υπάρχει ένα, ένας κίνδυνος ε, d'un gouvernement de juges λέει ο δηλαδή για μια κυβέρνηση δικαστών που θα επιβάλλει τι αποφάσει τη και βάσει αυτών θα κυβερνώνται οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι μια καλή σύμβαση η σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όμως οι πολιτικέ ερμηνείε κάποιων διατάξεων θα πρέπει να μην μα κάνουν να οδηγηθούμε σε ένα δημοκρατικό έλλειμμα και είναι θέματα αυτά τα οποία θα ήθελα να απευθύνω στους δικαστές. Ευχαριστώ. Είναι νομίζω ευκολότερο να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις μαζί οι ομιλητές μας. Ο κύριος Χένρι Λαμπάλη τώρα θα πάρει το λόγο. Εδώ είμαι πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις ε, θα κάνω, μάλλον δύο-τρεις ερωτήσεις. Ο Ζανκλόντ Μπονισό ε, μίλησε πολύ προσεκτικά για το ρόλο του δικαστηρίου ως προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σωστά είπε πως ε, το δικαστήριο ε, δεν έχει ως αποστολή να δικάζει επί των θεμελιωδών ε, ελευθεριών. Ε, ουσιαστικά δικάζει για συνταγματικά ή διοικητικά ζητήματα. Δίκαιο έχει. Ακούγοντας ε, τις επόμενες παρεμβάσεις όμως άρχισα να προβληματίζομαι, διότι από ό,τι κατάλαβα μας παρουσιάζεται το ε, σύστημα του Στρασβούρου και προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν ως τέλειο. Ε, Παρ' αυτά ε, δυσλειτουργεί ορισμένες φορές και δημιουργεί δυσκολίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τελικά πότε θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δικό της δικαστή για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί το ρωτάω αυτό διότι αδίκως ε, για πολύ καιρό σκεφτόμασταν ε, ιεραρχικά, σκεφτόμασταν ε, την, το διαχωρισμό των εξουσιών. Σήμερα αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν για αυτό το ζήτημα γιατί είναι προϋπόθεση για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχουν ναι, αυτόματα πολλαπλή ε, ε, Τα εθνικά νότατα δικαιοδοτικά όργανα, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Δεν πρόκειται πλέον για διελκυστίνδα ή για ε, παιχνίδι ισχύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σωστά είπε ο κ. Μπονισό, Α μην προσπαθούμε να οργανώσουμε την αταξία. Μα δεν είναι αυτό. Πρέπει να οργανώσουμε αυτή την πολυπολικότητα που διαπιστώνουμε, βρίσκοντας τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε εν ευθύνο, ευθέτω χρόνο ο καθένας μας να εκπληρώσει το ρόλο του για τον σεβασμό ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. παρότι κάποιοι αιρετοί ε, δείχνουν να θέλουν να ε, υποχωρήσουν σε σχέση με κάποιες δυσμεύσει τους. Αυτό στο οποίο αποσκοπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ε, μεγιστοποίηση τη συνεργασία ανάμεσα στα δικαιοδοτικά όργανα. Το θέμα των προδικαστικών ερωτημάτων προϋπήρχε του ενωσιακού δικαίου. Ήταν ένα ε, ένα μέσο που ε, επέτρεπε την ε, διαφύλαξη των αρμοδιοτήτων. Δηλαδή δεν μπορεί να επιλαμβάνονται μια υπόθεση ταυτόχρονα δύο δικαστές. Και στη συνέχεια μετατράπηκε σε μέσο συνεργασίας δύο δικαστών το προδικαστικό ερώτημα. Μία από τις βασικές προκλήσεις σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου και θα ήθελα την άποψη των αγορητών, είναι η εξής. Να οργανώσουμε και να θεσπίσουμε αυτό το διάλογο με αποτελεσματικό τρόπο και σε πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων όλων και προς ικανοποίηση όλων. Δεύτερη ερώτηση, ε, το θέμα της εξωεδαφικότητας. Θα επανέλθω και στην Τρογγύλη Τράπεζα αύριο σε αυτό το ζήτημα. Είναι λίγο αποκαλυπτικό το ζήτημα της εξοεδαφικότητα ε, για την ε, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εφαρμογή του χάρτη. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, θέτει κέρια, κέρια ερωτήματα, ε, δηλαδή ε, ζωή, θάνατος, βασανιστήρια, μου, αυτό είναι η εξοδαφικότητα. Οι περιπολία στην ανοιχτή θάλασσα, που βλέπουν ναι, σκάφη γεμάτα με παράνομους μετανάστες. Ε, λοιπόν, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο σε αυτή την περίπτωση. Ποιος θα εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων. Στο χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης λοιπόν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σήμερα να έχει ένα μοντέλο ε, που θα τύχει κοινή αποδοχή από όλα τα κράτη-μέλη. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, ε, η χάρτα προσφέρει περισσότερες αναλεκτικές λύσεις από ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, σωστά, ε, έχουν, οι αλλοδαποί έχουν προστατευτεί σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Αλλά όχι σε όλες τις ε, περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις σιώπησε το δικαστήριο του Στρασβούργου. Παραδείγματο χάρη σε περιπτώσεις πολιτικών προσφύγων ή όταν ε, πρόκειται για μέλη της ε, ε, οικογένειας του ετούντος άσυλο που βρίσκονται στην Καμπούλα ας πούμε. Ε, ταυτόχρονα, πέρα από τις επιπρόσθετες συναλλακτικές λύσεις υπάρχουν και σοβαρότεροι περιορισμοί μέσα στη χάρτα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Τέλος πάντων, για να κλείσω τι παρατηρήσει μου, δεν είμαι σίγουρο ότι το ίδιο πνεύμα διαπνέει τις εργασίες αφενός του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και αφετέρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστηρίο του Στρασβούργου του Λουξεμβούργου έχει κάνει επαναστατικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Μιλήσατε για την δυναμικότητα της ερμηνείας των ουσιαστικών δικαιωμάτων όπως ισχύουν σήμερα. Πρόκειται λοιπόν για εντελώς ε, διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ε, σε σχέση με το δικαστήριο που προσπαθεί ναι ε, να ε, προστατεύσει το πνεύμα των συνθήκων αλλά τελειολογικώς πώς ερμηνεύει το περιεχόμενο των συνθήκων και άρα το δικαστήριο του Στρασβούργου επειδή έπρεπε υπερεύει το, τη δράση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μπορεσό, οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Ο κύριος Σκίνερ. Από το γραφείο της Ethics for Europe στη Σουηδία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ το Ethics for Europe, μια μη κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί δέκα άλλε μη κυβερνητικέ οργανώσει από όλη την Ευρώπη. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε μια συγκεκριμένη περιοχή τη χάρτα που, που χρειάζεται προσωθυνισμό. Μιλήσατε, Πρόεδρε, ανοίγοντα την ακρόαση για τι προοπτικέ τη εφαρμογή τη χάρτα, ιδίω τη διαμόρφωση τη εθνική νομοθεσία στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο ήθελα να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για ένα συγκεκριμένο δικαίωμα που θεσπίζεται από το άρθρο 12, την ελευθερία του συνενώνεστε. Και ιδίως από την αρνητική πλευρά. Ενώ προβλέπει το δικαίωμα αυτό ο χάρτης, όπως και τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα της ε, σύμβασης, εδώ προβλέπεται η θεμελιώδης ελευθερία του συνεταιρίζεστε και της σύναψή ε, συμφωνιών. Έχει όμως καταστεί σαφέ ότι εδώ υπάρχει και το αντίθετο του, δικαιωμάτου, του δικαιώματος αυτού, το οποίο προκύπτει από την ομολογία του ΔΕΚ και είναι και κάτι που συζητήθηκε και στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου. Ένα βουλευτή το προηγούμενο τρίμηνο είπε ότι για να μπορεί να απολάβει το δικαιωμάτων του ένα άτομο, του δικαιώματο συγκεκριμένα του συνεταιρίζεστε, πρέπει να έχει και το δικαίωμα εάν θέλει να μην το κάνει. Εάν δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει και το άλλο. Καταλαβαίνουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη η εθνική νομοθεσία απαγορεύει την άσκηση της αρνητικής ελευθερίας. Και μα ανησυχούν κάποιες καταστάσεις στην Ευρώπη όπου ομάδες μειονότητα είναι θύματα διακριτική μεταχείρισης. Διότι αυτή η πτυχή της αρνητική ελευθερίας έχει παραμεληθεί. Το ερώτημά μου λοιπόν δεν αφορά τόσο το θεσμικό χαρακτήρα όλων των δικαστηρίων που ακουραστήκαμε και που πέρασαν σε πολλές λεπτομέρειες. Απλώς χαίρομαι που οι συμμετέχοντες του πάνελ είναι εδώ σε ειδικοί στα θέματα τους. Και επειδή η Επιτροπή ΛΥΜΠ υποδέχεται την εκδήλωση αυτή, θα έπρεπε να το εξετάσουμε αυτό νομίζω σε βάθο, σε συνεργασία ίσω και με την Επιτροπή των Αναφορών. Και να γίνει και μία δήλωση επί του θέματο που να καταγραφεί στα επίσημα πρακτικά τη ακρόαση. Και θα θέλαμε οι δυνατόν και συμμετέχοντες στο πάνελ να μπορέσουν να σχολιάσουν αυτό το σημαντικό θέμα και το πώ μπορεί να παραμελούνται αυτά τα αρνητικά δικαιώματα κάποιων ομάδων μειονοτικών. Ευχαριστώ. Η αντιπροσωπεία της Μερκοσούρ με μέλη από το Κοινοβούλιο της Παραγουάης θα ήθελα να θέσουν κάποια ερωτήματα. Τρία συγκεκριμένα μέλη από το Κοινοβούλιο της Παραγουάης. Ο κύριος Μπακίνη πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την, ε, το Κοινοβούλιο, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Μερκοσούρ και πιο συγκεκριμένα την ε, Παραγουάη. στο κοινοβούλιο μας μελετούμε ακριβώς αυτό το θέμα της συγκρότησης πρώτα απ' όλα ενός δικαστηρίου αρμοδίου για αυτά τα ζητήματα γιατί έτσι τα ψηφίσματα του Εθνικού μας Κοινοβουλίου θα γίνονταν ε, δεσμευτικά για, όλα τα, για όλες τις χώρες μέλη του Μερκοσούρ. Συνεργαζόμαστε στενά ε, με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Eurolat κάθε εξάμεινο έχουμε την κοινή συνέλευση ε, και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, όπου εκπροσωπούνται όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, όχι μόνο οι χώρες μέλη του Μερκοσούρ. Οι σχέσεις μας ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ε, επιτρέπουν να αντλήσουμε διδάγματα από τις δικές σας εμπειρίες ούτως ώστε με τη σειρά μας ε, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ταχύτερα αυτήν την υπερεθνική λύση, δηλαδή ε, την συγκρότηση ενός δικαστηρίου για το Μερκοσούρ. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ, Πρόεδρε, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε Ευχαριστούμε και όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Κύριος Σάλλη, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε να επανέλθουμε ε, στο αμερικανικό σύστημα προστασίας ε, των δικαιωμάτων ε, αυτός ο οργανισμός για όλα τα ε, κράτη της ε, Αμερικανικής Υπηρού εδρεύει στην ε, Ουάσιγκτον. Επιθυμεί δε αυτός ο οργανισμός να δημιουργήσει μια υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα εξετάζει τις υποθέσεις παρεμβαίνει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες μέλη του Μέρκοσούρ και γενικότερα στη Λατινική Αμερική. Οι πολίτες του Μερκοσούρ με πλέον ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο θα την χάνουν πλέον ε, προστασίας ε, ως προστευασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσει που έγιναν σήμερα εδώ, κυρίως για τα δικαιοδοτικά θέματα, πιο συγκεκριμένα ε, μιλώντας για τη δυνατότητα προσφυγής, άμεσης προσφυγής από πλευράς ε, των πολιτών σε αυτήν την υποεπιτροπή στην Ουάσιγκτον. Συζητούμε ήδη την κοινοβουλευτική συνέλευση του Μερκοσούρ αυτό το θέμα, διότι εξετάζουμε την δυνατότητα ίδρυσης ε, μονίμου δικαιοδοτικού οργάνου ε, σε επίπεδο Μερκοσούρ που θα επιφορτιστεί με την εξέταση των υποθέσεων παραβίασης των κανόνων του Μερκοσούρ, δηλαδή ένα όργανο αντίστοιχο προς το δικαστήριο του Λουξεμβούργου το Δικαστηρίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κάποια αντίσταση βέβαια από πλευράς ε, των ε, μεγαλύτερων χωρών, των ε, πλέον σημαντικών χωρών, δηλαδή της Αργεντινής και της Βραζιλίας, που δεν βλέπουν ευμενώς αυτή την ιδέα συγκρότησης του σώματος σε επίπεδο Μερκοσούρ. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου του Μερκοσούρ εξετάζει τώρα αυτό το θέμα, αλλά ακόμη δεν έχει καταδειχθεί είναι βιώσιμη η πρόταση. Και η διάσκεψη των Προέδρων των χωρών του Μερκοσούρ ούτω ή άλλω δεν έχουν εξετάσει ακόμη αυτή την ιδέα και δεν έχουν τοποθετηθεί. σω όμω ε, να σε ενδιαφέρει αυτή η ιδέα και γι' αυτό και την αναφέρουμε. Η συγκρότηση ενός τέτοιου δικαιοδοτικού οργάνου ε, προσφέρει ε, νομική ασφάλεια και θα προσφέρει νομική ασφάλεια σε χώρε που προσχωρήσουν ε, στο Μερκόσουρ. Ευχαριστούμε. κύριος Κανίζη, τελευταία παρέμβαση συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοι, παρακολουθήσαμε ιδιαίτερη προσοχή την ακρόαση αυτή για τις επιπτώσεις της εφαρμογής της χάρτας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι αυτού του είδους προσέγγιση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα θα επηρεάσει κατά τη διαδικασία... ευρωπαϊκής ολοκληρωσής, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Και εμείς, που η ανάλογη διαδικασία μας είναι πιο πρόσφατη, έχουμε θεσπίσει ίδρυση δικαστηρίου για να ασχολείται με εμπορικά και οικονομικά ζητήματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα Είναι ένα ζήτημα που το εξετάζει η Επιτροπή Αμερικανικών Κρατών. Όμως νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να σκεφτούμε εάν και αυτό είναι κάτι που έχει απασχολήσει τη Μερκοσούρ, να δούμε εάν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να εξετάσει περιπτώσεις ε, σύγκρουσης δικαιοδοσιών. Ένα δικαστήριο δηλαδή στο οποίο μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες. Ίσως θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε βάσει των ευρωπαϊκών σας εμπειριών. Eh, να μας στείλετε συμβουλές για το ποιος είναι ο δικαστικός χώρος στον οποίο θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Και τώρα να γυρίσω στους συμμετέχοντες, τους προσκεκλημένους μας, να σας παρακαλέσω να απαντήσετε στα ερωτήματα και στις παρατηρήσεις. Με τη σειρά που είχατε, ζητήσει, που είχατε παρέμβει και στην αρχική συζήτηση. Ο κύριος Μπονισό. Ας απαντήσω για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και την ε, αντιστροφή της Εάν μου επιτρέπετε θα απαντήσω στα γαλλικά γιατί για μένα είναι πιο απλό. και θα είναι και πιο ευχάριστο για εσάς. Για το ερώτημα αυτό να κάνω μια προκαταρκτική παρατήρηση γιατί είναι ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλές σε μένα. Εφόσον είμαστε και στο Ευρωκοινοβούλιο, να παρατηρήσω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Όσο περισσότερο εργάζεται στα θέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν σοβαρέ διαφορέ όταν μπαίνουμε στι λεπτομέρειε των δικαστικών συστημάτων, των δικαστικών παραδόσεων των επιμέρου κρατών μελών. Ε, από μακριά από απόσταση λέμε ότι τα συστήματά μα λίγο πολύ είναι οικοδομημένα στι ίδιες βάσεις και λογικά υπάρχουν πολλέ ομοιότητε. όμω όταν μπαίνει κανεί στι ε, λεπτομέρειες τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα, οι λεπτομέρειε είναι εξαιρετικά πολύ αριθμές, οι διαφορέ μάλλον, και έτσι είναι δύσκολο να καταλήξει κανεί σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τώρα για τον τομέα τη ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Δύο παρατηρήσει. Πρώτον, σε γενικέ γραμμέ ο τομέα αυτό αυτό καθεαυτό δεν είναι ο χώρος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες τις κοινοτικέ. Επαναλαμβάνει αγγλικά ο μιλητή. Κανονικά δεν εμπίπτει στι αρμοδιότητε τη κοινοτική, τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Όμω είναι προφανέ ότι μπορεί να υπάρξουν ε, παρεμβολέ εδώ, λόγω χάρη στον κοινωνικό τομέα. Όταν το δικαστήριο επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης όπου συζητούμε για, την υποχρεωτική, για τον υποχρεωτικό συνεταιρισμό την υποχρεωτική συμβολή των ε, εργαζομένων ή μισθωτών σε έναν οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ή όταν τα κείμενα θεσπίζουν την ίδρυση ένωσης αγροτικής, βιομηχανικής, όπου όλοι είναι υποχρεωμένοι να προσχωρήσουν. Στα πλαίσια μάλιστα μιας κοινή πολιτική. Το πρόβλημα προ στιγμήν και εντό των κοινοτικών νομοθετήτων δεν έχει τεθεί. Ενώπιον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάστηκε λόγω χάρη η γαλλική νομοθεσία στα θέματα του κυνηγιού. Όπω ξέρετε, είναι κανεί υποχρεωμένο να έχει συμμετάσχει σε συγκεκριμένου συλλόγου κυνηγών προκειμένου να μπορεί να κυνηγήσει στη Γαλλία. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι ναι, το πρόβλημα αποκλείται να τεθεί. Μπορεί να τεθεί. Μπορεί να τεθεί και στο κοινοτικό κεκτημένο, αλλά προ στιγμήν, εξ όσων εγώ γνωρίζω, δεν έχουμε σχετική νομολογία χαρακτηριστική αυτή τη κατηγορία των ε, αποφάσεων των δικαστικών που έχει εκδώσει λόγω χάρη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου. Και μια παρατήρηση εν παρόδο, Πρόεδρε, για την οικονομική ολοκλήρωση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων ελευθεριών, όπως τις έθιξαν ε, μόλις τώρα οι βουλευτές της Παραγουάης. Η όλη ιστορία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος δείχνει ότι τα δύο ζητήματα αυτά είναι τελείως αλληλένδετα. Ευτής εξ αρχή τέθηκαν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πρώτη απόφαση που το ΔΕΚ τοποθετήθηκε το θέματα αυτά είναι η Ρεφ Στάουμπερ του 1969. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δηλαδή, αλλά όταν βγει κανείς εκτός του οικονομικού χώρου. Και αυτό αναγκαστικά θα συμβεί, όχι μόνο για πολιτικούς λόγους. Τότε αναγκαστικά εξακολουθεί να οδεύει τον δρόμο τη οικονομική ανάπτυξη, αλλά είναι αδύνατο ταυτόχρονα να μην καλύψει τα δικαιώματα των πολιτών και των ε, προσωπικών και δημόσιων ελευθεριών. Όταν μιλάμε λοιπόν για πολιτική ολοκλήρωση και εφόσον θέλουμε να χτίσουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε και το ξέρει ακόμα περισσότερο από όλου ε, εδώ το Ευρωκοινοβούλιο, τον χώρο ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Πώ να γίνει αυτό χωρί να μιλάμε για δημόσιε ελευθερίε, για την ελεύθερη κυκλοφορία, των ατόμων. Πώς να υπάρξει κοινή πολιτική μετανάστευσης χωρίς να ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προφανές νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά είναι αλληλεξαρτώμενα. Ευχαριστούμε κύριε Μερχιόρ. Ε, ένα ερώτημα που ίσως δεν απευθυνόταν ε, αποκλειστικά σε μένα, αλλά να πω ότι εδώ έχουμε μια τούρτα λίγο πολύ. Δηλαδή τη θεωρία της κυβέρνησης, των δικαστών, οι οποίοι θα υποκαταστήσουν τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού. Πράγματι, κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει μια τάση να δημιουργείται τέτοια κυβερνητική εξουσία στα χέρια των δικαστών όταν υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους οι δικαστές τις, δικα... τις αρμοδιότητες για τις οποίες διορίστηκαν. Όμως το να φροντίζει κανείς το σεβασμό των ε, νόμων Αυτό σημαίνει ότι φροντίζει κανείς και την προστασία όσων ήταν υπέρ ενός τέτοιου κανόνα, ενός δικαιώματος δηλαδή, αλλά μετά μπορεί να υπάρξει και ακύρωση αυτής της απόφασης και αυτό βέσω δικαστικής απόφασης η οποία θα είναι πλήρως τεκμεριωμένη. Τώρα για την εξοδαφικότητα. Εάν ε, θυμηθούμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα δικαιώματα που καλύπτει η Σύμβαση αναγνωρίζονται στα άτομα που εμπίπτουν εντός της δικαιοδοσίας των συμβαλωμένων μερών. Όλα δηλαδή έχουν να κάνουν με το εύρος της δικαιοδοσίας της κάθε χώρας των συμβαλωμένων μερών. Πότε θα έχουμε ένα κοινοτικό δικαστή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μα υπάρχει, υπάρχει, αλλά δεν είναι ο πρώτο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όμως εξ αφορμής τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωσης το δικαστήριο του Λουξεμβούργου θα επαγρυπνεί Ήδη το κάνει, αλλά θα το εντείνει. Θα επαγρυπνεί λοιπόν για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση. Πραγματικά είναι μια ουσιώδης ερώτηση ο συσχετισμό μεταξύ νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας και αν εδώ υπάρχουν κάποια όρια τα οποία τα ξεπερνάμε, υπερβαίνουμε τα εσκαμμένα ή όχι. Θα έλεγα το εξή: πάντα όταν είναι συμβαλόμενο μέρος ένα κράτο, τότε υπάρχει περιορισμός των κυριαρχικών του δικαιωμάτων κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι τόσο σαφέστερο φυσικά όταν έχουμε και ένα δικαστήριο το οποίο επιτηρεί κάποια πράγματα και κάποια, ε, κάποιες Ένα δικαστήριο το οποίο σε συγκεκριμένα θέματα μέσα στη δικαιοδοσία του παραμένει και νομολογεί. Παρόλα αυτά πρέπει να πούμε όμως ότι πάντα υπάρχει ένα πεδίο έντασης μεταξύ αυτού που αρχικά ήθελαν οι ιδρυτές των συνθήκων και αυτού που μετεξελίσσεται στη συνέχεια μέσω διαρκούς νομολογίας ε, και δραστηριότητας δικαστικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να αναφέρω και ένα άλλο σημείο. Εδώ έχουμε για παράδειγμα την ε, ε, παρουσίαση ε, από πλευράς του Βρετανού δικαστού που στην παρέμβασή του το 2009 τι ανέφερε ήταν αποχαιρετιστήριος λόγος του και είπε ότι καμιά φορά συνέβαινε στα θέματα αυτά της νομολογίας του 10 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να υπάρχει αυτή η διτή τροχία και πράγματι αυτή είναι η απάντησή μου εδώ. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τη στοχοθέτηση του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ε, δικαστηρίου στο ε, Μόναχο για παράδειγμα. Το ε, πρέπει να μεριμνά να ε, προχωρά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι σε σχέση με θέματα ερμηνείας ε, δεν υπερβαίνουν καμιά φορά τα εσκαμμένα όσον αφορά τους αρχικούς στόχους. Είναι όμως ένας θεμητός στόχος αυτός, γιατί ουσιαστικά πρόκειται και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο μόλις προανέφερα, όταν είχαμε το θέμα της αυστηρής ερμηνείας του άρθρου 51. Δηλαδή το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο να εφαρμόζεται, διότι διαφορετικά θα υπάρχουν στρεβλώσεις και ακριβώς είναι έργο του δικαστηρίου να αποφευθούν οι στρεβλώσεις ε, και οι καταχρήσεις. Όσον αφορά τις άλλες παρεμβάσεις που έγιναν, θα ήθελα να αναφερθώ ως εξής. Θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου και εγώ στην φωνή του δικαστού Μπονισό και όσον αφορά την παρέμβασή του θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλες παρεμβάσεις παρακαλώ. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτών των δύο γύρων παρεμβάσεων. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τις ε, προτάσεις, παρεμβάσεις και για τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είδαμε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα, πόσο ενδιαφέρουσες είναι οι πτυχές αυτές και πόσα μπορούμε να κερδίσουμε, να αποκομίσουμε για τις μελλοντικές συζητήσεις ε, αναγνωρίζοντας ε, το εύρος και το πλούσιο πεδίο αυτών των λεπτομεριών. Έχουμε ευρύ πεδίο. Θα συνεχίσουμε αύριο λοιπόν στις 9 με τη συνεδρίαση για την ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια, χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα δούμε και τον, τους πανεπιστημιακούς, τον ακαδημαϊκό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών. Θα έχουμε τον την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ρέντινγκ, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, κύριο Κύρον. Θα έχουμε ε, επί, αντιπρόσωπο από την ε, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Απλά και μόνο θα ήθελα να αναφέρω για αύριο το πρώτο τμήμα της πρωινής ε, συνεδρίασης με αυτά τα λόγια. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και τις παρεμβάσεις σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.